Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της απογευματινής μας συνεδρίασης. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά περιμέναμε τον κύριο Άγγλη μέχρι τώρα που ακόμη όμως δεν εμφανίστηκε. Περνάμε σε ένα πολύ ευχάριστο θέμα, την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Γεωργίας της Εστονίας, τον κύριο Τάρμο Τάμ, ασκώντα την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα γεωργίας. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, καλωσορίζουμε τον εκπρόσωπο της Εστονικής Προεδρίας. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η δυνατότητα αυτή για συζήτηση μαζί σας. Θυμόμαστε την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε στο Αγκροφόρουμ για τη Βαλτική, το Αγκροφόρουμ Mare Balticum. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν τα προβλήματα της γεωργίας στην Ευρώπη και θα θυμάστε τη συνάντηση που είχατε με την, Επιτροπή, με την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας. Μάλιστα είχαμε και ξεχωριστή συνεδρίαση των συντονιστών μας μαζί σας. Οπότε είχαμε την ευκαιρία για μια σύντομη ενημέρωση επί των προτεραιοτήτων της Εστονικής Προεδρίας. Τώρα θα γίνει μια πιο διεξοδική παρουσίαση του προγράμματος της Εστονικής Προεδρίας σε θέματα γεωργίας. και κατόπιν ε, θα δώσω το λόγο στους συντονιστές και μετά στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ε, καλωσορίζω φυσικά και το επιτελείο σας, τους συνεργάτες σας και τους βουλευτές που, ήταν, που δεν ήταν στην πρωινή συνάντηση. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Σικέρσκη και εσείς συντονιστές των πολιτικών ομάδων και ευρωβουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας για να σας εξηγήσω τις προτεραιότητες της πρώτης εστονικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξα βουλευτής στο Εστονικό Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια και βλέπω με μεγάλη ικανοποίηση την αύξηση της επιρροής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά πράγματα γιατί αυτό αποτελεί ένα σημάδι δύναμης ευρωστίας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της δυνατότητας να μεταφέρεται καθαρά η φωνή των ε, ψηφοφόρων στο επίπεδο της Ένωσης. Η Εστονία είναι μικρή χώρα, περίπου όσο η Ολλανδία, με πληθυσμό όμως μόλις 1,3 εκατομμύρια κατοίκων. Ως μικρή ανοιχτή χώρα η ασφάλεια και η ευημερία μας εξαρτώνται από την ικανότητά μας να αποτελέσουμε μέρος μεγαλύτερων ομάδων που μοιράζονται τα ιδανικά μας. Πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για την Εσονία κορυφώθηκε η προσπάθεια αυτή με την ένταξή μας πρώτα 13 ετών, μας έκανε όμως πιο ισχυρούς και πιο, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μία από τις θετικές πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η πολυφωνία και το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη τις γνώμες των μικρών χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει πολλά στην Εστονία. Με την Προεδρία μας ελπίζουμε να ανταποδώσουμε. Πριν προχωρήσω στην εισαγωγή των, του προγράμματος εργασιών μας, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα την Προεδρία της Μάλτας που προηγήθηκε και που μπορούμε να βασιστούμε στο έργο μας για να προχωρήσουμε, στο έργο της, συγγνώμη, για να προχωρήσουμε. Τα κύρια καθήκοντα, αποστολές της ε, Προεδρίας μας θα είναι να συνεχίσουμε την πορεία της νομοθετικής ολοκλήρωσης και της λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο. Εκπροσωπούμε εξάλλου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα. Η ε, διαδικασία συναπόφασης σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό ρόλο αποφασιστικής σημασίας. Εξ αυτού του λόγου είμαι ακόμα πιο ικανοποιημένος που βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα, ενώπιον δηλαδή της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου. Για μας είστε σημαντικός εταίρος. Πιστεύω σε μια θετική συνεργασία μεταξύ μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων το επόμενο εξάμεινο σύνθημα της Προεδρίας μας είναι ενότητα μέσω της ισορροπίας. Η Εστονία πιστεύει στην ενότητα της Ευρώπης και έχουμε το στόχο να επιτύχουμε εξισορρόπηση δυνάμεων για την επίτευξη λύσεων. Οι προτεραιότητες μας θα είναι πρώτα μια ανοιχτή καινοτόμως ευρωπαϊκή οικονομία με προώθηση των θεμελιωδών ελευθεριών και την απλούστευση των οικονομικών δραστηριοτήτων με διαμεθοριακό χαρακτήρα. Μια Ευρώπη ασφαλή που θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για την κρίση το μεταναστευτικό και να ενισχύσουμε την εσωτερική ασφάλεια. Ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να θα συνεχίσουμε μάλλον την προσπάθεια να κρατήσουμε ανοιχτές τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες και θα προωθήσουμε την ελεύθερη διακίνηση δεδομένων και επιγραμμικών υπηρεσιών. Ε, σε αυτά η Ιστονία παίζει πρωτοπόρο ρόλο στην Ευρώπη. Θέλουμε μια ανοιχτή Ευρώπη που να περιλαμβάνει στους κόλπους της όλους. Αξιότιμα μέλη και εσείς κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω με τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας μας στον τομέα της γεωργίας. Εκεί θα ρίξουμε το βάρος μας στον εξυγχρονισμό και απλούστευση της κοινή αγροτική πολιτικής και στον κανονισμό Omnibus. Θα σας μιλήσω επίσης για ζητήματα διεθνούς εμπορίου. Η κατάσταση στις αγορές των αγροτικών προϊόντων, την προστασία των γεωργικών γεών, τον αγώνα κατά της αντίστασης στα ε, αντιβιωτικά και βεβαίω θα μιλήσω και για την σημασία της προστασία των ζώων αλλά και της υγεία φυτών και ζώων. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι μειώνονται οι πόροι, από την άλλη μεριά αυξάνεται η ζήτηση για τρόφιμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία. Θεμέλιος λίθος των οικονομικών πολιτικών της Ένωσης αποτελεί μεταξύ άλλων και η γεωργία. Πρέπει να συνεχιστεί η κοινή αγροτική πολιτική για να στηρίζει την γεωργία και την ανάπτυξή της. Οι συζητήσει για το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική έχουν ήδη ξεκινήσει και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο Υπουργών. Και είναι ουσιώδου σημασία αυτό και ω θέμα προτεραιότητα τη Προεδρία μα. Ο Το έγγραφο προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δημοσιονομικά που δημοσιεύθηκε ε, αρχές Ιουλίου δεν αποτελεί την καλύτερη βάση. Τέσσερα από τα πέντε σενάρια προβλέπουν μείωση του προϋπολογισμού. Αυτό, ε, κάτι τέτοιο, θα σημάνει μεγαλύτερη πίεση και ανάγκη ανάληψης ευθυνών από τον αγροτικό τομέα. Αποτελεί πρόκληση βέβαια για, το, για τις συζητήσεις για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Έχουμε τώρα τα αποτελέσματα της ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης για τον εξυγχρονισμό της κοινή αγροτικής πολιτικής που αποτελούν σημαντική εισρωή, σημαντικό input για το μέλλον της ε, κοινή αγροτικής πολιτικής. Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα ήταν ότι η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει ενιαία πολιτική, κοινή πολιτική. Όμως ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι χρειάζεται εξυγχρονισμό και απλούστευση. Ταυτόχρονα σημειώνεται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες της κοινωνίας και των γεωργών σε ό,τι αφορά την ε, έκβαση της πολιτικής αυτής. Η εξέβρεση ισορροπίας ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η Εστονία θα συνεχίσει την πορεία των προηγούμενων προεδριών για την κατεύθυνση που θα δίνει δηλαδή στις συζητήσεις για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Θέμα το οποίο θα απασχολήσει το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας θα διεξαχθεί στο Ταλίν τον Σεπτέμβριο. Λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια των βασικών γεωργικών αγορών των τελευταίων ετών και λαμβάνοντα υπόψη και την ανάγκη καλύτερη προετοιμασία για τι προκλήσει του μέλλοντο καθώ και του δημοσιονομικού περιορισμού, ε, θέλουμε εμεί να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε μέτρα διαχείριση των κινδύνων στη μελλοντική ΚΑΠ. Γνωρίζω ότι στην Επιτροπή σα έχετε διαξαγάγει σε βάθο συζητήσει για το θέμα αυτό. Κύριε Σικιάσκη, για σας μάλλον θέλω να πω ότι αναμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι συζητήσεις μας στο Ταλίν. Σε ό,τι αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, για μα η απλούστευση εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Προτεραιότητά μα είναι να προχωρήσουμε γρήγορα τον κανονισμό Omnibus με στόχο να επιτύχουμε διοργανική συμφωνία το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα θα ρίξουμε το βάρος μας στις πτυχές εκείνες που συμβάλλουν σε μια πραγματική απλούστευση των όρων και διατάξεων της κοινή αγροτικής πολιτικής. Θεωρώ ότι εκεί θα παίξετε εσείς ένα σημαντικό ρόλο και είμαι πεπισμένος ότι η συνεργασία μας θα συνεχιστεί καρποφόρα τους επόμενους μήνες. Στη διάρκεια της Εστονικής Προεδρίας θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε δει σημαντικές διακυμάνσεις και κρίσεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια και ιδίως στα γαλακτοκοπικά, οποροκυπευτικά και στο χείριο κρέας. Ακόμα και σήμερα αισθανόμαστε τους αντικτύπους του ρωσικού εμπάργου σε ορισμένους τομείς γεωργικών προϊόντων. Και αυτό χαρακτηρίζεται και από την επέκταση των ιδιαίτερων μέτρων, των ειδικών μέτρων δηλαδή, σε ορισμένους τομείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως Προεδρία είμαστε διατεθειμένοι να αντιδρούμε στις διακυμάνεις αυτές των ε, αγορών θέτοντας τα θέματα προς συζήτηση. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς αποδίδουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ενίσχυση της θέσης των παραγωγών μέσα στη, στην αλυσίδα ε, παροχής προμήθειας τροφίμων. Χρειάζεται να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και στις διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές αγροτικών προϊόντων. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την νομοθετική πρωτοβουλία καλύτερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από τα πιο σημαντικά εξαγώγημα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και τα ποτά. Ο τομέας αυτός παίζει σημαντικό ρόλο και στην δημιουργία απασχόλησης στον αγροτικό τομέα. Χρειάζονται λοιπόν ξεκάθαροι κανόνες για την παραγωγή και για τις επενδύσεις. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για ε, τον κανονισμό, για την νομοθεσία δηλαδή, στον ε, τομέα των υνοπνευματοδών ε, ποτών. Όσον αφορά το έργο οργανώσεων διεθνών οργανώσεων, εμείς εκεί θέλουμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε σημαντικό να διατηρήσουμε πολιτικές ανοιχτού εμπορίου και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να συνάψουμε εμπορικές συμφωνίες που να ωφελούν τον αγροτικό τομέα της Ένωσης. Αυτό θα διευκολύνει τους Ευρωπαίους παραγωγούς να ανοίξουν νέες αγορές. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σώμεθα και εμείς υπέρ της αρχής της διαφάνειας στα θέματα αυτά. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνει τακτικά τις χώρες μέλη για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων διεθνών και πολυμερών για εμπορικές συμφωνίες. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας θα οργανώσουμε μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου με στόχο να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή για την βιώσιμη χρήση των γεών, διότι γόνιμα εδάφη είναι κέρια για το μέλλον της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πάνω από 95% της ποσότητας αλλά και της ποιότητας των καθημερινών μας, αυτό που καθημερινά βρίσκουμε στο πιάτο μας εξαρτάται από την ποιότητα των εδαφών. Το μέλλον της ανθρωπότητας εξαρτάται από το τι συμβαίνει στα 20 πρώτα εκατοστά των ε, στρωμάτων των εδαφών. Θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε ιδιαίτερα την σημαντική αυτή πρόκληση για την διατήρηση της ποιότητας των γεωργικών γεών. Γνωρίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί ενεργά το θέμα αυτό και αναμένω συνεργασία μαζί σας προς την κατεύθυνση αυτή. Η Εστονία πιστεύει ότι ο παγκόσμιος αγώνας κατά της αντίστασης κατά των αντιβιωτικών έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς συμβάλλουμε για την εφαρμογή της One Health Policy που ισχύει για ανθρώπους, φυτά και ζώα. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον δημοσίευσε σχέδιο το οποίο συζητήθηκε τον Ιούλιο στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλίας. Εμείς θα οργανώσουμε και ε, διάσκεψη για το θέμα της μικροβιακής αντοχής τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες για να προωθήσουμε τα θέματα του One Action Health ε, Plan Σε ό,τι αφορά την νομοθεσία, θα συνεχίσουμε την εργασία μας και με αντικείμενο ε, τα σχέδια νομοθεσίας για ε, ζωοτροφές που περιέχουν αντιβιωτικά και ούτω καθεξής, οι δε τεχνικές συζητήσεις του Συμβουλίου έχουν προχωρήσει. Θα προωθήσουμε τις αναγκαίες συμβιβαστικές λύσεις, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με χορήγηση διαπραγματευτική εντολή πριν από το τέλος της Προεδρίας μας. Θέλω να τονίσω επίσης την σημασία της προστασία της υγεία των ζώων και των φυτών και για τη γεωρική παραγωγή αλλά και γενικότερα προ όφελο της κοινωνία. Τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα και τους αξίζει ο σεβασμός μας. Είναι σημαντική η συμβολή στον τομέα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόσφατη πλατφόρμα υγεία των ζώων αποτελεί το σωστό φόρουμ για να συμμετάσχουν όλα τα μέρη σε ανταλλαγή απόψεων και να συντονίσουν το έργο τους. Ως Προεδρία στηρίζουμε και αν χρειαστεί συμπληρώνουμε τις δραστηριότητες του φόρουμ, της πλατφόρμας, με νομοθετικές προτάσεις για την βελτίωση της προστασίας των ζώων με εθελοντικές δεσμεύσεις. Η κατάσταση στις μολυσματικές ζωονόσους χρειάζεται διαρκή προσοχή εκ μέρους μας. Το Συμβούλιο συζητεί τα θέματα αυτά τακτικά. Αποδίδουμε μεγάλη αξία στην συνεργασία των ελέγχων των ζωονόσων μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις χώρες μέλη και τρίτες χώρες. Στον φυτογειονομικό τομέα η Εστονία θα συνεχίσει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης, όπως ξεκίνησε η Προεδρία της Μάλτας, θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη σχεδιασμών για αντιμετώπιση επιουσών καταστάσεων, για να είμαστε έτοιμοι και προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε ξέσπασμα ε, ζωονόσου. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η ψηφιακή Ευρώπη για μας. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας και μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουμε διάσκεψη για συστήματα διαχείρισης πληροφοριών που φέρει τα αγγλικά αρχικά IMSAC. Θα στηρίξουμε συζητήσεις που θα επιτρέψουν στις χώρες μέλη να αρχίσουν να χρησιμοποιούν σύγχρονες ψηφιακές λύσεις για την εφαρμογή μέτρων ελέγχου. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, μόλις σας έκανα μια σύντομη παρουσίαση των στόχων της Προεδρίας μας. Τόνισα τις βασικότερες προτεραιότητές μας. Το πιο σημαντικό θέμα, ωστόσο για μας, είναι η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η επίτευξη συμφωνίας για τον κανονισμό Omnibus και βεβαίως για το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής. Θα παρακολουθούμε άλλωστε προσεκτικά τι εξελίξεις στις αγορές αγροτικών προϊόντων και απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στηρεί τακτικά ενήμερους για τις διεθνείς και για πολυμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα επίσης στα θέματα της ανθεκτικότητας των εδαφών. Η μικροβιακή αντοχή επίσης είναι προτεραιότητα για μας. Θέλουμε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή, δηλαδή με συζητήσει για καλύτερα φάρμακα, κτηνιατρικά και φαρμακούχες ζωοτροφές. Και με εταίρους εσά, τα άλλα θεσμικά όργανα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι πρόθυμος να ακούσω τις προτάσεις και τις συστάσεις σας, συστάσεις και στη σημερινή συζήτηση, αλλά βεβαίως και στο μέλλον. Ελπίζω δε η συνεργασία μας στο επόμενο εξάμεινο να αποδειχθεί κακοφόρα. Επιθυμώ να σε ευχαριστήσω και πάλι που με προσκαλέσατε να εμφανιστώ ενώπιόν σας και θεωρώ ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να ελπίζουμε σε μια πολύ κακοφόρο και γόνιμη συνεργασία τους επόμενους έξι μήνες. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ. Όπως σας είχα υποσχεθεί και προηγουμένως, ε, περνάμε στη συζήτηση. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές και και πρώτα απ' όλα τον συντονιστή του ΕΛΚ, τον κύριο Ντες. Ο κύριος Ντες, ευχαριστώ πολύ και σας κύριε Υπουργέ και σας κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Τάρμο, χαίρομαι που μετά το γεύμα είστε παρόν εδώ ενώπιόν μας στην Επιτροπή Γεωργίας Βλέπω τη σημασία αποδίδεται στην εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλωστε και εσείς υπήρξατε για πολλά χρόνια βουλευτής. Είπατε ότι η Εστονία είναι μικρή χώρα. Ωστόσο, έχω μια προσωπική εμπορία, μια προσωπική εμπειρία. Αποχαιρετήσαμε την σωρό του Helmut Kohl. Το 2004, όταν έφυγα από τη Γερμανική Βουλή και ήρθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πήγα και αποχαιρέτησα προσωπικά τον Helmut Kohl, τον οποίο γνώριζα προσωπικά πολύ καλά. Και μου είπε, φεύγοντα, κάτι το οποίο θέλω να σου το αποκαλύψω. Μου είπε, ασχολήσου όταν θα πά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τι μικρέ χώρε, γιατί χωρί τι μικρέ χώρε δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν το μήνυμα του Helmut Kohl και ήθελα να σα το μεταφέρω και σήμερα εδώ. Παρουσιάσετε το πρόγραμμα της ε, Προεδρίας σας. Χαίρομαι πολύ που αναλαμβάνετε την Προεδρία γιατί είμαι βέβαιος ότι υπό την ηγεσία σας θα προχωρήσουμε πολύ στον γεωργικό τομέα. Ήδη κάναμε μια πρώτη συνάντηση μαζί με τον Πάολο Ντεκάστρο για τον κανονισμό Omnibus, γιατί ο Πάολο ήταν εισηγητής. Είδαμε λοιπόν ότι η Εσθονική Προεδρία προσέρχεται στις συνομιλίες αυτές καλά προετοιμασμένη και με διάθεση να συνεργαστεί. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο και που το λέγω ως εισηγητής εδώ του Κοινοβουλίου, θέλω να μπορέσουμε να προωθήσουμε στο συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που έχουμε τον, τη συζήτηση για τον κανονισμό Omnibus. Να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τον Οκτώβριο. Θα πρέπει να περάσουμε τα θέματα το ένα μετά το άλλο. Σημαντικό είναι βέβαια το Συμβούλιο Υπουργών να καταλήξει σε θέση. Δεν είναι απλό για σας βέβαια να καταφέρετε να αποκτήσει κοινή θέση το Συμβούλιο το είδαμε για παράδειγμα στην κοινή οργάνωση, στις κοινέ οργανώσεις αγοράς ότι το Συμβούλιο δεν έχει καταφέρει να τοποθετηθεί. Δεν φταίτε εσείς διότι εσείς μόλις 1η Ιουλίου αναλάβατε την ευθύνη. Αλλά χρειαζόμαστε θέσεις του Συμβουλίου για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Είπατε ακόμη ότι είναι σημαντική η στήριξη των παραγωγών. Συζητήσαμε τα πράγματα αυτά σήμερα το πρωί. Πράγματι εδώ τη συζήτηση για τον κανονισμό έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το δυνατόν συντομότερο νομοθετικές προτάσεις, διότι εδώ χρειάζεται ανάληψη δράσης. Επιτρέψτε μου να τονίσω, ξαναλέω, όταν το 2004 έγινε για πρώτη φορά Ευρωβουλευτής, αρχίσαμε την συζήτηση περί περιαγωγής και πριν από λίγες μέρες καταργήθηκαν τελείως τα τέλη περιαγωγή. χωρί νομοθετικέ προτάσει από την Ευρώπη, τα τέλη περιαγωγή θα ίσχυαν ακόμα στην κινητή τηλεφωνία. Να λοιπόν που αποδεικνύεται η ανάγκη ότι χρειάζονται νομοθετικέ πρωτοβουλίε. Και για την ενίσχυση τη θέση των γεωργών χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία. Από τη μια μεριά είναι η μεγάλη πολυεθνικοί όμιλοι που παράγουν γεωργικά προϊόντα, από την άλλη είναι η παραγωγή που χρειάζεται ενίσχυση την θέση τους, η θέση τους. Σε ό,τι αφορά τι εμπορικές συμφωνίες, πρέπει να προσέξουμε, να λαμβάνονται υπόψη τα γεωργικά συμφέροντα. Συμφωνίε με Νέα Ζηλανδία, με Αυστραλία που επίκειται, Μερκοσούρ, άλλο όπου πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερη, να ρίξουμε ιδιαίτερη έμφαση. Και σα υπενθυμίζω κύριε Υπουργέ ότι το 2010 και τελειώνω αποφασίσαμε στο Συμβούλιο ότι οι εισαγωγέ γεωργικών προϊόντων από τρίτε χώρε θα επιτρέπονται μόνο εφόσον γίνονται σεβαστέ οι προδιαγραφέ μα για προστασία καταναλωτών, φυτών και ζώων. Αυτό πρέπει να έχει προτεραιότητα ακόμη σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι και μένουμε με μεγάλη χαρά την συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστούμε. Επειδή είχαμε μιλήσει προηγουμένως στη συνεδρίαση των συντονιστών και είχαν ήδη ξεσπάσει και είχαν μιλήσει αρκετά. Ήλπιζα οι συντονιστέ να μην χρειάζονται τόσο χρόνο. Αλλά εδώ είδα ότι όχι μόνο δεν τήρησαν το δίληπτο, αλλά μακρηγόρησε και όλο ο κύριο πρώτα. Ο κύριο Αντρέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω και να σα καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή Γεωργία, κύριε Υπουργέ. Ήταν πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψε που είχαμε και στο Τάρτου, στο Αγκροφόρουμ. Και βλέπουμε πόσο πλούσιο είναι το πρόγραμμα της Εστονικής Προεδρίας αυτού του εξαμήνου και σίγουρα θα είναι πολύ σημαντική επιτυχία και κρίσιμη για το μέλλον της Γεωργίας. Μιλήσατε φυσικά για την κοινή γεωργική πολιτική, για την απλούστευση, την απαιτούμενη. Το είπαμε και το πρωί. Σίγουρα η μελλοντική αναθεώρηση ε, εντάσσεται σε πολύ περιορισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επειδή κάθε μέρα μιλάμε για τον Brexit, δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό το θέμα τώρα. Πάντως, ε, χαρακτηρίζει τις δημοσιονομικές, ε, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οπότε θα πρέπει αυτό το θέμα να το λάβει το Συμβούλιο στο επόμενο εξάμεινο. Και με βάση τη μελέτη που έγινε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη να δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη μελλοντική αναθεώρηση. Μα είπε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στα τέλη του έτου θα υποβάλει την ανακοίνωσή τη ή στι αρχέ του επόμενου έτου. Οπότε θα πρέπει όλοι από κοινού να δώσουμε κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ ή κάποιο προσανατολισμό. Εσεί ε, μα είπατε ακροθυγώ ποιο μοντέλο προ το οποίο θέλετε να προσανατολίσετε τη μελλοντική μεταρρύθμιση. Είναι μικρή χώρα μεν η Εστονία, αλλά μα ενδιαφέρει γιατί οι οικογενειακέ εκμεταλλεύσει ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι οι πιο πολυάριθμε. Οπότε και το θέμα της ποιότητα τροφίμων και το θέμα τη προστασία ε, του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία θέσης απασχόληση και τη προστασία του εδάφου, σχετίζονται άμεσα και με τι ε, μικρέ αυτέ οικογενειακές εκμεταλλεύσει. Επίση, μιλήσατε για την εμπορική πολιτική. Έχουμε ενώπιό μα πολύ σημαντικέ διαπραγματεύσει. Το Μερκοσούρ είναι ήδη εδώ. Ναι. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσει ε, ήδη με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για εμπορικέ συμφωνίε και ξέρουμε ότι τα γεωργικά ζητήματα θα είναι πολύ σημαντικά και σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Οπότε θα πρέπει να μεριμνούμε και να επαγρυπνούμε γενικώ ε, για το πώς θα η υπόψη η γεωργία σε τέτοιου είδους εμπορικές συμφωνίες. Επίσης, ε, η ύψιστη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι ο κανονισμός Omnibus. Ευχαριστώ που το αναφέρατε και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας για τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ποιότητα των εδαφών. Μίζων πρόκληση η ποιότητα του εδάφους και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και γενικώ. και θα πρέπει να προβληματιστούμε στο ύψιστο δυνατό επίπεδο με το θέμα της ποιότητας των εδαφών. Συγχαρητήρια λοιπόν για την πρωτοβουλία σας, τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ποιότητα των εδαφών, γιατί πραγματικά το θέμα μας απασχολεί Σε Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Τα βιολογικά είναι εκτός ε, συζήτηση, οπότε θα γλιτώσετε τη συζήτηση σε σχέση με σε αντίστοιχα με τους προκατόχους. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που είχατε να πείτε, αλλά θυμάμαι την προηγούμενη μετάρρυθμιση της ΚΑΠΑ και ακούω τα ίδια επιχειρήματα κατά του προπολισμού Γεωργία, ότι είναι πολύ μεγάλο, ότι θα πρέπει να περικοπεί κτλ. Ο προηγούμενο ομιλητή αναφέρθηκε σε διάφορα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο προπολογισμό, όχι μόνο στη χώρα μου. Και επειδή θα φύγουμε από την Ένωση, δεν θα ήθελα να δω διακρίσει κατά των υπολείπων Ευρωπαίων Γεωργών. και πρέπει να σας αναφέρω την σημασία του προπολογισμού τους επόμενους μήνες. Γιατί αν δεν έχουμε τα κονδύλια τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Εμείς προσωπούμε μια βιομηχανία. Εσείς αναφερθήκατε ας πούμε στα, στα ρωσικά αντίμετρα. Δεν ξέρουμε λοιπόν πότε θα συμβεί το επόμενο πρόβλημα, η επόμενη καταστροφή, το επόμενο πρόβλημα στον προστατολισμό της αγοράς. Και αυτό βέβαια είναι πολύ καλό, πολύ κακό συγγνώμη για τους καταναλωτές και για τους γεωργούς. Πρέπει να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε. Και είδαμε τις ενδεχομένες λύσεις που είχαμε μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να μάθουμε από όλα αυτά. Και νομίζω ότι η ΚΑΠ αποτελεί μια μεγαλύτερε προκλήσεις μαζί με αυτά που αναφέρατε προηγουμένως. Και κάτι άλλο. Πέρσι στην Ευρώπη πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι πλωρικών αντιμετώπισαν προβλήματα όχι μόνο λόγω υγείας ε, λόγω γρήβης των πτηνών. Αλλά είχαμε μεγάλη οικονομική καταστροφή για πολλούς λόγους για αυτούς τους κτηνοτρόφους. Τώρα έχουμε φτάσει σε, σε ένα σημείο όπου δεν ξέρουμε τι γίνεται και βέβαια δεν θέλω να συμβεί αλλά Ανησυχώ πάρα πολύ που δεν έχουν υπάρξει συζητήσει, κουβέντε, δεν έχει γίνει τίποτα για το συγκεκριμένο ζήτημα από τότε που έχει ανακύψει. Και αυτό νομίζω αφορά πολλούς άλλους τομεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τα σχόλια του κυρίου Νίκολσον για τον προϋπολογισμό. Ε, ήταν πραγματικά εύστοχο το επιχείρημα και να μην ξεχνούμε ότι για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2014-2020 ε, ε, ο γεωργικός προϋπολογισμός ήταν κατά 11% λιγότερο, 38 ε, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσιονομική περίοδο, με τις προηγούμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Ήδη έχει μειωθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός. Και αυτή η μείωση κατά 11% ίσως είναι πολύ σημαντικό επιχείρημα. Θα πρέπει να το επικαλεστούμε γιατί έτσι θα είμαστε σε καλύτερη θέση στη συζήτηση. Κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ. που δηλώσατε ότι από διταξία στη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην συζήτηση μαζί μας η υγεία των ζώων όπως και η μικροβιακή αντοχή είναι πολύ σημαντικά πράγματα αλλά βέβαια και η παραγωγή πρωτεϊνών και η προστασία των εδαφών. Το σημαντικότερο εργοτάξιο θα είναι πραγματικά η ψήφιση του κανονισμού Omnibus και η επίτευξη πλειοψηφία. Και όχι μόνο εσείς στο Συμβούλιο Υπουργών έχετε ποικίλε γνώμε και απόψει, αλλά και εδώ στην Επιτροπή Γεωργία βεβαίω εκπροσωπούνται διάφορα ρεύματα. Έχω να σα πω μόνο ότι η θέση του κόμματός μου, της ΑΛΔΕ, των φιλελευθέρων δηλαδή, λέει καθαρά ότι έχει καλώσει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντως χρειαζόμαστε απλούστευση των διαδικασιών το δυνατόν ταχύτερα για τους Γιώργους, αλλά στεκόμεθα και πολύ κριτικά απέναντι στις ε, προτάσεις για, την, ε, για, τους, για τις οργανώσεις των αγορών οργανώσεις παραγωγών, οργανώσεις ε, καταναλωτών, όλοι αυτοί πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά τι περιλαμβάνει το πακέτο των γαλακτοκομικών και πού ακριβώς εντοπίζονται τα προβλήματα. Όταν γνωρίζω ότι 3,5% μπορεί να, ε, να δημιουργηθεί ως δέσμη από την πλευρά λοιπόν των παραγωγών, ε, υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα εκεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Εάν τώρα αυτό είναι ο σωστό τρόπος, δεν θέλω να το αξιολογήσω προσωρινά. Γεγονός είναι πάντως ότι στην Γερμανία απέναντι στο προηγούμενο χρόνο έχουμε παραδόσεις κατά 2% λιγότερων ποσοτήτων γάλακτο. Το ίδιο σημαίνει και στη Γαλλία, 3,5%. Παρόλο που δεν διοχετεύεται χρήμα στην αγορά αυτή. Το, η τιμή του βουτύρου έχει ανέβει. Πρέπει να φροντίσουμε ο παραγωγός μας ο οποίο λειτουργεί ω επιχειρηματίας να μπορεί να αντιδράσει στις εξελίξει αυτές. Προσέξτε λοιπόν αυτές τις οργανώσεις αγορών. Εμείς των φιλελευθέρων θεωρούμε ότι αυτά που έχουμε ως μέτρα αρκούν για την ώρα και δεν μπορούμε να παίρνουμε μονομένα προβλήματα με μονομένων χωρών που έχουν ελλείψει στις δομές τους να τα βάζουμε στο μεγάλο αυτό πακέτο. Δεν θέλουμε καινούρια κοινή αγροτική πολιτική, θέλουμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας πραγματικά στα απαραίτητα, δηλαδή στην ουσία σε αυτή τη γραφειοκρατική απλούστευση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χόισλινγκ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είπατε πολλά για αυτά που θέλετε να προωθήσετε. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε πράγματι με τον κανονισμό περί βιολογικών. Χρειάζεται να κάνετε τις τελευταίες πινελιές. Τα βασικά προβλήματα τα έχουμε ήδη λύσει. Αλλά ελπίζω η οικολογική γεωργία να είναι σημαντική και για σας. Και για τη χώρα σας άλλωστε είναι σημαντικός οικονομικός τομέας. Και βέβαια πρέπει να ασχοληθούμε τώρα με την κοινή αγροτική πολιτική, δεν το αμφισβητώ αυτό. Θα Πρέπει όμως ε, να ξεφύγουμε από την ιδέα ότι πρέπει να παραμείνουν τα πράγματα όπως είναι. Πρέπει να ακούσουμε τι λένε και οι 350.000 πολίτες οι οποίοι συμμετέσχουν στη διαβούλευση. Χωρίς την υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών που είναι ψηφοφόροι αλλά και φορολογούμενοι δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα. Πράγματι υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε πολλά στην κοινή αγροτική πολιτική. Δεν αρκεί όμω να πούμε ότι μειώνουμε τη γραφειοκρατία, αλλάζουμε τι προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε εάν ο προσανατολισμός του πρώτου πυλώνα πραγματικά εξακολουθεί να είναι χρήσιμη, χρήσιμο εργαλείο. Άλλοι μίλησαν εδώ για τα ζητήματα του Διεθνού εμπορίου. Ασκήσαμε και τη σχετική κριτική. Το ίδιο για τι διαπραγματεύσει με τις χώρες Μερκοσούρ, το ίδιο για τις χώρες Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία. Μας λείπει η διαφάνεια. Εμείς ως ενδιαφερόμενοι και που επιμένουμε στην προστασία των συμφερόντων μας ως γεωργοί και ως παραγωγή, περιμένουμε και περιμένουμε και δεν βλέπουμε να γίνεται τίποτα. Έχουμε και εμείς οι ευρωβουλευτές το δικαίωμα να ζητήσουμε διαφάνεια. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε απλά να μας θέση υπόψη εν τέλει ένα κείμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κείμενο συμφωνίας ενώ το οποίο απλώ προσυπογράφουμε ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσφατη συμφωνία με την Ιαπωνία. Σωστά μιλήσατε και για την προστασία των γεωργικών γεών και μιλήσατε και για διάσκεψη. Είμαι απόλυτα σύμφωνος. Πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο όντως οφείλουμε να δώσουμε ιδιαίτερο ε, ιδιαίτερη έμφαση. Πράγματι, πρόκειται για τα 20 πρώτα εκατοστά του εδάφους, τα οποία εξασφαλίζουν σε όλη την ανθρωπότητα το προστοζήν. Πρέπει να προσέξετε επίσης όμως κάτι που θέλουμε να προωθήσουμε με νέα έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ζήτημα της παραγωγής λευκομάτων, πρωτεϊνών δηλαδή. Η εξάρτησή μα από τι εισαγόμενε πρωτεΐνες είναι πολύ υψηλή. Χρειαζόμαστε στρατηγική παραγωγής πρωτεϊνών. Μιλήσατε και για την προστασία των φυτών. Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους μου εδώ που λένε ότι για την προστασία τους χρειάζεται νέα προϊόντα της χημίας, θεωρώ ότι πρωτίστως πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των αντιστάσεων στα διάφορα μικροβιοκτώνα, ζενιοκτώνα κλπ. Και όχι να επιτρέπουμε όλο και να εγκρίνουμε όλο και περισσότερα προϊόντα. Χρειάζεται λοιπόν μια νέα στρατηγική και όχι μοναχά αδειοδότηση όλο και νέων ε, σκευασμάτων. Ευχαριστώ κύριο Σουλαζό. Ευχαριστώ πρόεδρε την Κομισιόν για την απλούστευση της ΚΑΠ. Πράγματι το συζητάω εδώ και καιρό. Επιτόπου όμω δεν έχει συμβεί τίποτα. Εξάλλου αντιστέκονται οι Γεωργοί επειδή ξέρετε ότι έχουμε πολλού ελεγχού και ξέρω τι εννοώ γιατί και εγώ ίδιο είμαι Γεωργό, κύριε Υπουργέ. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον αγώνα δρόμο για εξαγωγέ, Αντί να δούμε προτεραιότητα στα προϊόντα μα και να αναπτύξουμε τι δικέ μα επιχειρήσει για να αντισταθούμε στι εισαγωγέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους ε, συντονιστές. Περνάμε στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ο κύριος Δεκάστρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω πραγματικά τον Υπουργό Τάμα και την Εστονική Προεδρία. Όπω είπε ο Στάναφος έχουμε εμπιστοσύνη. Είχαμε ήδη ένα πρώτο τριμερή διάλογο για το Omnibus. Και νομίζω ότι για κάποια σημεία του Omnibus, όπως έχει κινδύνου που αναφέρατε, ξέρω ότι αυτά είναι θέματα που η Ιστονική Προεδρία προσέχει ιδιαίτερα. Και αυτό είναι και ένα από τα τρία μεγάλα κεφάλαια του Omnibus εξάλλου. Ήθελα λοιπόν εγώ στην παρέμβασή μου να τονίσω τη σημασία που έχει η επίτευξη κοινή θέση στο Συμβούλιο για την πλειοψηφία των διαφόρων θεμάτων. Επειδή είδαμε στον τριμερή διάλογο ότι η κοινή θέση δεν υπάρχει και αντιμετωπίσαμε δυσκολίες και μιας και ο χρόνος περιορίζεται θα έχουμε δύο τριμερείς βέβαια το Σεπτέμβριο, αλλά στην πράξη θα πρέπει να κλείσουν τα πάντα μέχρι τον Οκτώβριο. Οπότε εύχομαι να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου και να κάνουμε βήμα, προ, βήματα πρόοδου, χρησιμοποιώντας ακόμα και το άτυπο συμβούλιο. Ευχαριστώ. Α, παρακαλώ. Ο, ο χρόνος που χρησιμοποιήσει ο κ. Δεκάστρο είναι παράδειγμα προς μίμηση υπόδειγμα για όλους μας ο κύριος Δεκάστρο, τήρηση του χρόνου. Μας υπενθύμισε και τη διαδικασία με το Συμβούλιο. Ε, είχαμε την εμπειρία και από το κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα, πόσο δύσκολο ήταν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσει λόγω τη απροθυμία ε, του Συμβουλίου. Κύριο Κούσμιουκ, παρακαλώ, τηρήστε το χρόνο ομιλία που έχετε. Ευχαριστώ. έχω δύο ερωτήσει μόνο προ τον Υπουργό είπατε κύριε Υπουργέ για την αναμενόμενη περικοπή του γεωργικού ε, προϋπολογισμού για μετά το 2020. Και σίγουρα οι σχετικές ε, συζητήσεις θα ξεκινήσουν επί Προεδρίας. Ερωτώ, εσείς είστε υπέρμαχος τέτοιων περικοπών στο γεωργικό προϋπολογισμό. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα δημοσιονομικό κενό από το Brexit κανονικά θα πρέπει να χεβηρωθεί αυτό το κενό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Συμφωνείτε ή θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει να συμβάλλουν τα κράτη-μέλη για να γεμίσουν αυτό το δημοσιονομικό κενό, οπότε μας περιμένουν ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στο γεωργικό προϋπολογισμό, αν μείνουν αγεφύρωτα αυτά τα κενά. Επίσης, ε, είπατε ότι θα φροντίσετε να ενισχύσετε τη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα προμήθειας τροφίμων. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε τη διαπραγματευτική θέση των παραγωγών, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε επί της Προεδρίας γι' αυτό. Η συνεισφορά των κρατών μελών ε, για να γεφυρωθεί το δημοσιονομικό κενό είναι 15% ε, δηλαδή 23 δις περίπου. Βέβαια ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και με τις εκτός που λαμβάνει του επιστρέφονται κάποια ποσά. Οπότε ετησίως το δημοσιονομικό κενό είναι 11 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 4,5 δισεκατομμύρια λιγότερα το χρόνο έχουμε για τη γεωργική πολιτική. Επίσης, ε, στις συζητήσεις οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μένουν στο ποσοστό 15% και στα 23 δισεκατομμύρια. Δεν είναι όμως ακριβώς αυτά τα συγκεκριμένα ποσά, δεν είναι αυτό το δημοσιονομικό κενό, γιατί θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις εκπτώσεις, τις επιστροφές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε μένουν μόνο 11 δισεκατομμύρια. Κυρία Αγγιλέρα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε και συζητούμε τα θέματα που μας απασχολούν. Και θα ήθελα να πω ότι από αυτά που επισημάνατε και που είναι σημαντικά είναι καταρχήν η απλούστευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ήδη μάλιστα η Επιτροπή μας ε, με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε πρόταση για τον κανονισμό όμνιμπους. Ελπίζω να τη λάβετε υπόψη γιατί έτσι θα σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο. Και μια και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία δεν αναμένεται άλλη σημαντική μεταρρύθμιση, μάλλον η μεταρρύθμιση θα απασχολήσει την επόμενη κοινοβουλευτική θητεία, ελπίζω να λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας για τον κανονισμό Omnibus. Επίσης, το θέμα της ενίσχυσης των παραγωγών στην τροφική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι δύο επιτροποί, Χόγκαν και Βεστάγκερ, υποσχέθηκαν ότι θα υποβάλουν νομοθετική πρόταση για την επόμενη άνοιξη για αυτό το θέμα. Και στο μέτρο που και η Εστονική Προεδρία είναι υπέρ της πρωτοβουλίας, ελπίζω να προχωρήσει γρήγορα, γιατί συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση της θέσης του παραγωγού στην τροφική αλυσίδα. Πολύ χρήσιμη ήταν και η πρωτοβουλία του Επιτρόπου Ανδριουκάητης για την ενιαία υγεία, One Health, και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής. Επ' αυτό θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή μας συζήτησε επί της ουσίας το θέμα των φαρμακούχων ζωοτροφών. Δεν μπορούμε όμως να ξεκινήσουμε παράλληλα τον τριμερή διάλογο και για τα κτηνιατρικά φάρμακα, γιατί η αρμόδια κατ' ουσία για αυτό είναι η Επιτροπή Έμβη, ε, είμαστε για τα, τις φαρμακούχες ζωτροφές, Αλλά πολλά θέματα από το κυρίως ζήτημα θα πρέπει να διεκπαιρεωθούν πριν περάσουμε στο επόμενο. Οπότε καλό θα ήταν στο δικό σας εξάμεινο να προωθήσετε τον τριμερή διάλογο για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς λίγους μήνες μετά να ξεκινήσουμε τον τριμερή διάλογο για τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Επίσης, Πολύ σημαντικό είναι και το θέμα των αλκοολούχων ποτών, όπω είπατε. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη τι πρακτικέ των κρατών μελών και τι εθνικέ νομοθετικέ διατάξει. Αν δεν λάβουμε υπόψη την εθνική νομοθεσία στον κανονισμό για τα αλκοολούχα ποτά, ίσω οδηγήσουμε στον αφανισμό σημαντικέ παραδόσει και προϊόντα που έχουν μακραίωνη παράδοση. Είναι κρίμα λοιπόν να χάσουμε τέτοια προϊόντα. Λάβετε παρακαλώ υπόψη τι εθνικέ νομοθεσίε. Σα ευχαριστώ κυρία Χόιμπουχ. Äh, Ευχαριστώ πολύ και εσά κύριε Πρόεδρε και εσά κύριε Υπουργέ. Δύο θέματα με απασχολούν που ω τώρα δεν ακούστηκαν. Αφενό η συγκέντρωση των έδαφων. Εξακολουθούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου 80% των ενισχύσεων της κοινή αγροτικής πολιτικής πηγαίνουν σε 20% των εκμεταλλεύσεων. Αυτό οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση εδαφών. Ενώ αρχικά η ΚΑΠ είχε ως στόχο να ενισχύσει όλες τις ιωικές εκμεταλλεύσεις και να εξασφαλίσει τη ζωή και των μικρών. Το Κοινοβούλιο έχει εγκύψει στον προβληματισμό αυτό. Ερώτηση τώρα, κατά πόσον εσείς και η Εστονία θα μας υποστηρίξετε. Χρειαζόμαστε καλύτερη δικτύωση μεταξύ των χωρών μελών για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει και υπερεθνικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, τι ε, σκέπτεστε για την ιδέα να γίνονται τακτικά τεχνικές συναντήσεις, οι χώρες μέλη να συνεννοούνται μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις σε τεχνικό επίπεδο και να προσφέρουν υποστήριξη μεν στις δε. Δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να μας υποστηρίξετε ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας καλύτερα δεδομένα για βελτιωμένο monitoring για την συγκέντρωση γεών στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάνουμε προσπάθειες να συλλέξουμε στατιστικά δεδομένα. Τα πράγματα αυτά πρέπει να γίνουν με μεγαλύτερη διαφάνεια. Να γνωρίζουμε όταν γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι αποτελούν μέρος ενός διεθνούς ομίλου. Εκεί είναι πολύ δυσδιάκριτες οι δομές και δεν γνωρίζουμε εν τέλει και πού διοχετεύονται τα χρήματα της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας είναι η μικροβιακή αντοχή. Είπατε ότι κάνετε ένα σχεδιασμό. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με τα αντιβιωτικά τα οποία ε, κατευθύνονται, ε, χρησιμοποιούνται για την υγεία των ανθρώπων και χρησιμοποιούνται και στις κτηνοτροφικές μονάδες. Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκεται η συζήτηση. Η συγκέντρωση των γεών ε, έχει και κάποια θετικά αποτελέσματα περισσότερη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, με καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αλλά αυτό αφορά κυρίως το εξωτερικό εμπόριο. Υπάρχουν δηλαδή και υπέρ και κατά. Εγώ συμφωνώ μαζί σας βέβαια. υπάρχουν περισσότερα μειονεκτήματα από τη συγκέντρωση γεών παρά πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποιες θετικές πτυχές και αυτή είναι η τάση προς τη συγκέντρωση γεών, γιατί επικρατεί η οικονομική πτυχή. Ο κύριος Δενανό καταφτάνει ο, ο Υπουργό σε μια σημαντική στιγμή για την προετοιμασία της μελλοντική ΚΑΠ. Τι να σας πω, σα άκουσα, αλλά <laughs> δεν ξέρω τι να πω γιατί ζητάμε εδώ και πολύ καιρό την απλούστευση και τα άκουσα τώρα το πότε επιτέλου. Πάντω. έχουμε τα θέματα του περιβάλλοντος, Έχουμε το θέμα της αστάθειας των τιμών, της αξιομοιώσης. Δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιήσετε τεχνικές, ας πούμε, που θα επιτρέψουν να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Να σας ρωτήσω, γιατί έχω αναλάβει μια έκθεση για τις παρθενίνες; τι άποψη έχετε για τις αντισταθμίσεις στα φυτικά στα φυτικά ελλείμματα στην Ένωση, δηλαδή αύξηση της παραγωγής των πρωτεϊνών. Γιατί εδώ πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και βεβαίως να προχωρήσουμε και η χρήση των δαφών. Νομίζω ότι υπάρχει μια καλή πρωτοβουλία για μια συνάντηση στο Τάλιν. Ελπίζω να συμμετέχουμε πολλοί από εμά γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για την βιωσιμότητα. Και να καταλήξω λέγοντας μην ξεχνάτε και το θέμα της ψηλής ταχύτητας για τους γεωργούς. Χρειάζεται ψηλή ταχύτητα στους η ευρυζωνικότητα του ίντερνετ για τους γεωργούς είναι απαραίτητη σήμερα για κάτω δουλειά τους. Σας ευχαριστώ κύριε Σουροπέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ καλή τύχη και καλή επιτυχία στην Εσθονική Προεδρία. Σας ευχαριστώ για το πρόγραμμά σας που το βρίσκω ιδιαίτερα φιλόδοξο. Και έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας και θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Αναφερθήκατε στην εξίσου των συνθηκών για τους γεωργούς που θα πρέπει να είναι ισότιμες από τη σκοπιά του ανταγωνισμού. Δεν αναφερθήκατε όμως στα καθεστώτα ενίσχυσης. Ποια είναι τα σχέδιά σας για τα καθεστώτα ενισχύσεων στο μέλλον, γιατί και σε αυτά έχουμε μεγάλες διαφορές και ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Οπότε αυτή η διαφορά στα καθεστώτα ενίσχυση επηρεάζει τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός με τέτοιες διαφορές. Επίσης, Αναφερθήκατε στην ενίσχυση του ρόλου των γεωργών και της διαπραγματευτικής τους ε, ισχύς, ε, ισχύως στις, ε, στην τροφική αλυσίδα. Πώς σκοπεύετε να το κάνετε. Βέβαια ένα εξάμεινο δεν αρκεί για εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά μπορείτε να δώσετε μια όθηση για την επόμενη Προεδρία και να, συνεχίσουν, να συνεχιστούν οι αγαστές προσπάθειες για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύω του γεωργού στην τροφική αλυσίδα. Θα πρέπει να διδαχθούμε και από τα παθήματα του παρελθόντος, δηλαδή την κρίση στη, στο γαλακτοκομικό τομέα και να προβλέψουμε ένα μηχανισμό διαχείρισης των κρίσεων, ώστε να μην χρειάζεται τελευταία στιγμή να επιλύουμε ε, άρον-άρον μία κρίση και να μας ευνηδιάζει, να μας πιάνει απροετοίμαστος θα πρέπει να είμαστε ήδη έτοιμοι για να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις, για να μην τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Επίσης, ε, να προβληθεί ένα καθεστώς ενίσχυσης των νέων γεωργών, ώστε μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά γεωργικών γεών. Στην Εστονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία έχουμε μεγάλο πρόβλημα με την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων. Σκοπεύετε να λάβετε κάποιο μέτρο, γιατί ε, και πλήττει ιδιαίτερα τους γεωργούς στις χώρες της Βαλτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που έθεξε ο κύριος Νίκολσον. Την γρήπη των ποινών. Και το πόσο έχει επηρεάσει και τους πτηνοτρόφους με κοτόπουλα ελεύθε, ελευθέρας βοσκής. Και μάλιστα η προθεσμία των 20 εβδομάδων ε, προβληματίζει και τους Ολλανδούς πτυνοτρόφους. Θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα η πρόταση. Μέχρι στιγμής μας έχει κοστίσει ε, σε άμεσες ε, ζημίες 10 εκατομμύρια ευρώ η γρήπη των πτηνών. Προσπάθησα να ζητήσω από τον Επίτροπο Χόγκα να βρει μια κατάλληλη λύση, αλλά ακόμη απάντηση δεν έχω πάρει. Σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της κρίση, τη γρήψη των πτηνών. Επίση, μιλήσαμε για το ρωσικό εμπάρκο. Στι 7 Αυγούστου του 2013 θυμάμαι την πρώτη μου συνεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πόσο συζητούσαμε την επιρροή του ρωσικού εμπάργου στους παραγωγούς προκυπευτικών τυριού, ε, χείριου κρέατος και ούτω καθεξής. Εσείς τι γνώμη έχετε, πώς μπορούμε να αναζητήσουμε μια καλή λύση για να αντιμετωπίσουμε το ρωσικό εμπάργο ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ. Τον Υπουργό για αυτά που μας είπε. Ήδη πολλές ερωτήσεις ακούστηκαν από τους υποβλήθηκαν από τους αδέλφους. Νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το μέλλον της ΚΑΠ και από το Brexit. Τα σε εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οπότε πιστεύω ότι πια ή θα πρέπει να αυξηθούν οι εισφορές των χωρών μελών ή θα έχουμε μειώσει στις δαπάνες. Οπότε οι κάποιοι άλλες πολιτικές όπως ε, κοινωνικές πολιτικές θα υποφέρουν πρώτες. Εσείς τι άποψη έχετε γι' αυτό. Θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε κάτι για την πολιτική συνοχή. Τι άποψη έχετε γι' αυτό. Μετά για τη συγκέντρωση των γεών αυτό είναι ένα μεγάλο φαινόμενο, αρνητικό και είναι δύσκολο να το ελέγξουμε. Δεν μπορούμε όμως να μην διαπιστώσουμε την ύπαρξη νομοθεσίας στις χώρες μέλη. Εμείς θεωρούμε ότι ας πούμε για την Ανατολική Ευρώπη κάποια πράγματα ισχύουν που δεν ισχύουν όμως σε άλλες χώρες μέλη. Σε κάποιες λοιπόν χώρες μέλη έχουμε κάποιες προϋποθέσεις. Παραβαίνει η Κομισιόν και υποχρεώνει την, την επιβολή της διαδικασίας επί παραβάση. Άλλες χώρες δεν αποδέχονται αυτή τη διαδικασία. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές θέσεις, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια κοινή θέση για όλες τις χώρες. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο πυλώνα, ο δεύτερος πυλώνας αφορά περισσότερο τον εξυγχρονισμό της γεωργίας. Και η μεταφορά κονδυλίων από το δεύτερο πυλώνα στη πολιτική συνοχή θα σήμαινε τεράστια απώλεια ε, για τη γεωργία. Βέβαια και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να, προσ... να βοηθά στη επίλυση των προβλημάτων το... της υπαίθρου. Ευχαριστώ κυρία Εράς Γκαρσία. Ε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η επιτυχία μια Προεδρία δεν έχει καμία σχέση με το μέγεθο τη χώρα που την ασκεί, αλλά είναι άμεση συνέπεια τη βούληση ε, υπέρ της ευρωπαϊκή ολοκλήρωση που έχει κάθε Προεδρία. Οπότε, αν ήταν επιτυχημένη η Μαλτέζικη Προεδρία, που επίση ήταν από μικρό κράτο, φαντάζομαι το επιτυχημένη θα είναι και η Εσθονική. Χαίρομαι που δίνεται σημασία στον κανονισμό Omnibus θα πρέπει να δώσουμε μια αόθηση στον κανονισμό αυτό στη διάρκεια τη Προεδρία σα Και ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο φιλόδοξο για τον κανονισμό Omnibus από ότι το Συμβούλιο. Ερωτώ λοιπόν, έχετε ήδη ένα πρόγραμμα δράσης για να μας βοηθήσετε και να συνεργαστούμε ώστε να προωθήσουμε τον κανονισμό Omnibus. Αναγγέλθηκε μια καθυστέρηση ό,τι αφορά τις νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Αυτό ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβετε κάποια δράση. Η Λετωνική Προεδρία λέει, κύριε Ράς. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριο Σάνι. Uh, ευχαριστώ, Υπουργέ να συμφωνήσω με αυτούς που μίλησαν θετικά για την παρέμβασή σας και για το σχέδιο της Προεδρίας σας. Αναφερθήκατε ιδιαίτερα στην καινοτομία και μιλήσατε για κάποιες προόδους στον τομέα της ψηφιοποίησης του ελέγχου στη Γεωργία. Κάτι το οποίο καλωσορίζω. Υπάρχει όμως ένα περαιτέρω βήμα και το θέτω προς εξέταση. Δηλαδή εδώ στο Κοινοβούλιο εργαζόμαστε πάνω σε μια πρωτοβουλία που ονομάζεται ΦΥΗ Χωριά και έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση στις περιοχές της και επικεντρώνεται στους κατοίκους της Υπέθρου πάνω από το 1 τρίτο δηλαδή του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Ένα ε, μεγάλο θέμα αυτό σημαντικό. Θα ήθελα τα σχόλια σας από αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλάνναγκαν. Ευχαριστώ. Λυπάμαι που καθυστέρησα γιατί μου σε άλλη συνεδρίαση και έχασα την εισαγωγική σας παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό Omnibus και την ευκαιρία που μας δίνει να κάνουμε κάτι για τους νέους γεωργούς ε, και να καταστήσουμε το σύστημα πιο ευέλικτο ώστε να μην εμποδίζουμε τους νέους ε, που θέλουν να ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα να το κάνουν ή όσοι έχουν ε, ε, εργαστεί ε, ως μερική απασχόληση με τη γεωργία στην οικογενική εκμετάλλευση και τώρα δεν είναι επιλέξιμη. Γι' αυτό καταθέσαμε τροπολογία στην, στον κανονισμό του Όμνιμπους για να συμπεριληφθούν και αυτοί. Εσείς πώς σκοπεύετε να διευκολύνετε τους νέους γεωργούς για την ανάληψη δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά το Natura 2000, δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα στην ιεραρχία ή κάπου αλλού. Πάντως εμείς έχουμε πρόβλημα στην Ιρλανδία με την εφαρμογή του Natura 2000. Ένας επιθεωρητής τους λέει να κάνουν το α, μετά διαβάζουν εγχειρίδια που τους λένε να κάνουν το β και υπάρχει πρόβλημα με την εφαρμογή του Natura 2000. Και πραγματικά δεν σας ζηλεύω καθόλου που πρέπει να απαντήσετε στις ε, ερωτήσεις, τόσο πολύ άριθμες, θα χρειάζεστε ένα πεντάωρο, αν θέλετε, να τις αντιμετωπίσετε όλες. Ο κύριος Γιάρ. Ε, ευχαριστώ και εγώ είχα χρειαστεί να ε, πάω σε άλλη ε, κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω τις εισαγωγικές σας τοποθετήσεις. Σας ευχαριστώ πάντως για την διάθεσή σας να απαντήσετε. Ε, βεβαίως θα μετρηθείτε σε αυτή τη διαδικασία του κανονισμού Omnibus συμπαρατάσσεστε περισσότερο με το Κοινοβούλιο ή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα είναι το πρώτο ερώτημα που θα σας θέσω. Δεύτερο, έχουμε εγκρίνει ορισμένα πράγματα ως Κοινοβούλιο και βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι έχουμε προβλέψει και την διαδικασία του κανονισμού Omnibus να παραταθεί η ισχύ ορισμένων διατάξεων, ιδίω διότι κάποια προγράμματα στον γεωργικό τομέα αρχίζουν να λειτουργούν τώρα και η επόμενη μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι από το 2020. Ε, πώς σας φαίνεται αυτή η παράταση, η χρονική παράταση. Και ε, μια τελευταία παρατήρηση. Στην διαδικασία του κανονισμού Omnibus περιλαμβάνουμε και κάποια στοιχεία από, γραφ, από ε, γραφειοκρατοποίησης. Ε, πώς σας φαίνονται οι ιδέες αυτές που προβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Δηλαδή μείωση της γραφειοκρατίας στην αγροτική μεταρρύθμιση, αν πρόκειται να τη στηρίξετε ή όχι. Όντως, η στόχοι του κανονισμού Omnibus παρά είναι φιλόδοξοι και μάλιστα προκαταλαμβάνουν κάποιες πτυχές της μεταρρύθμισης και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ξέρουμε πόσο δύσκολο θα είναι για την Εστονική Προεδρία να καταλήξει σε συνένεση σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική εντολή για τον κανονισμό αυτό. Κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο παρακαλώ. Σύντομα, Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλή τύχη με την Προεδρία σα Έμουν χθε το τάλι με τον Πρωθυπουργό σα Οπότε στερίζω τι προτεραιότητε τη προεδρία σα. Είδα τα σχολεία σας σε σχέση με την μακροβιακή αντοχή. Αφορά και άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή περιβάλλοντο είναι ένα σημείο κλειδί για μας. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για αυτό το θέμα και θα ήθελα να ακούσω λίγο περισσότερο για αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω τις ευχές μια καλή τύχη στην Προεδρία σας. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Α, μας, έλειψε στην αρχή ο κύριος Άγνιο. Έχετε το λόγο. Λυπάμαι και ζητώ συγγνώμη κύριε Υπουργέ. Είχα και εγώ άλλη συνεδρίαση. Πάντως σας είχα συναντήσει και το πρωί. Ε, δεν ξέρω αν κανένα μίλησε για τα φυτοφάρμακα. Γιατί φαίνεται ότι έχει κηρυχθεί πόλεμος κατά των φυτοφαρμάκων από το λόμπι των πρασίνων. Έχουμε τρία μέτωπα, ενδοκρινικούς διαταράκτες, την απαγόρευση για τα νεονικοτινοειδή, όχι μόνο στις ανθοφόρες καλλιέργειες για να προστατευτούν οι μέλισσες, μέλισσες αλλά και αλλού που δεν έχουμε επικονίαση από τις μέλισσες. Και, και το τρίτο μέτωπο είναι η γλυφοσάτη αν ε, οι πράσινοι κερδίσουν τι μάχε και στα τρία μέτωπα, θα μειωθεί η γεωργία. Οπότε θα αναγκαστούμε να εισάγουμε μαζικά γεωργικά προϊόντα από άλλα ε, μέρη του κόσμου και θα α, ε, είναι πολύ ευνοϊκή μεταχείριση των τρίτων χωρών σε σχέση με του δικού μα γεωργού που θα υποστούν αθέμητο ανταγωνισμό. Μάλιστα. Ήρθε η ώρα σας κύριε Υπουργέ για να απαντήσετε. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι είναι τιμή μου που είμαι εδώ σήμερα γιατί είμαι υπουργό από μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν, είναι και τόσο, δεν είμαστε και τόσο μικροί αν μα εγκρίνει κανεί με την Μάλτα. Και μια και η Μάλτα τα κατάφερε κατά διάρκεια τη, Προεδρία της, θα τα καταφέρουμε και εμεί Και συνεργασία με το Κοινοβούλιο αλλά και την Κομισιόν κατάφερε η Μάλτα να περάσει τον κανονισμό για τη βιολογική καλλιέργεια. Οπότε η Μάλτα μας έδειξε ότι μια μικρή χώρα μπορεί να καταφέρει πολλά με τη βοήθεια και των υπολείπων. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν όλους για τις ερωτήσεις σας. Βέβαια θα χρειαστούν πέντε ώρες να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά αν σας πειράζει θα τις ε, συμπτύξω σε θεματικές ενότητες. Ελπίζω να μην σας πειράξει, ε, έτσι, αν δεν υπάρξουν προσωπικές απαντήσεις, αλλά δεν έχουμε χρόνο και θα τις συνοψίσω όπως έλεγα. Καταρχάς, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι η μεταρρυθμίση η μελλοντική της ΚΑΠ. Οι συζητήσεις μόλις έχουν ξεκινήσει και θα θέλαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά των προηγούμενων προεδριών. Εμείς παρακολουθήσαμε τη συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για την μελλοντική κατεύθυνση της ΚΑΠ μετά το 2020. Βλέποντας λοιπόν το μέλλον της ΚΑΠ, Ελπίζω και τα δύο θεσμικά όργανα να μπορέσουν να συμφωνήσουν για το γεγονός ότι η αγροτική πολιτική θα πρέπει να παραμείνει κοινή πολιτική και ότι η κοινή αυτή η αγροτική πολιτική θα πρέπει να τυχαίνει εμπαρκούς οικονομικής στήριξης. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση με προσανατολισμό προς την αγορά. Θα πρέπει όμως να είναι και εύκολο να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική και να είναι σε θέση να αντισταθεί στις κρίσεις. Αναμένουμε βεβαίως την ανακοίνωση της Κομισιόν για το μέλλον της ΚΑΠ. Ελπίζουμε αυτό να γίνει σύντομα και τότε θα ετοιμαστούμε για περαιτέρω συζητήσει. Επίση στην Εστονία θεωρούμε ότι αυτέ οι υπηρεσίε που ακούσαμε να γίνεται λόγο ψηφιοποίηση στην Υπέδρα κτλ. θα συμβάλλουν ακριβώ στην επίτευξη αυτών των στόχων, επειδή θεωρούμε ότι αυτές οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους νέους γεωργούς και είναι πολύ σημαντικό επίσης για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους και να τους διατηρήσουμε στις περιοχές υπαίθρου. Τώρα, για τους ε, κινδύνους και δεχείς των κινδύνων σε σχέση με την κοινή πολιτική. Αν δούμε τι έγινε με τις κρίσεις στην ΚΑΠ, θα δούμε ότι θα πρέπει βέβαια να ενισχύσουμε την δυνατότητα παραγωγή των ε, Γεωργό και να τους βοηθήσουμε να ταπεξέρχονται σε αυτές τις κρίσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν όταν μιλάμε για το μέλλον της ΚΑΠ να μιλήσουμε για δικλείδες ασφαλείας και για μέτρα α, αντιμετώπισης κρίσεων ώστε το μέλλον της Γεωργίας να διαθέτει πιο αποτελεσματικά εργαλεία και να σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τις κρίσεις. Κατά διάρκεια λοιπόν της Προεδρίας μας θα έχουμε το Συμβούλιο Γεωργίας Αλίας όπου θα συζητήσουμε αυτά τα μέτρα και αυτό είναι το σχέδιό μας. Τώρα θα συζητήσω το θέμα ή θα αναφερθώ στο θέμα του κανονισμού του Omnibus. Θεωρώ ότι η απλούστευση της κοινή αγωγική πολιτικής και η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι ένας από τους κύριους στόχους και παραμένει ένας από αυτούς. Έχουν γίνει ήδη αρκετά για την απλούστευση της ΚΑΠ Υπάρχουν όμω πάντοτε περισσότερε δυνατότητε περαιτέρω απλούστευση, οποιασδήποτε πολιτική γενικότερα. Και αν δούμε ακριβώ αυτό το θέμα τη απλούστευση, βλέπουμε ότι ο κανονισμό Omnibus διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα σημαντικά για τα οποία συμφωνούν και το Κοινοβούλιο αλλά και η Προεδρία. Είναι αλήθεια ότι το Κοινοβούλιο νομίζω ότι σκέφτεται περισσότερο το μέλλον από την Κομισιόν. Και ελπίζω να συνεργαστούμε σωστά. Τώρα για τις πολλές προτάσεις που αφορούν το προσθενίσμα, τους παραγωγούς, τη κίνδυνο κτλ. Είμαι βέβαιος ότι μετά από συζητήσει που έχουμε σχεδιάσει να κάνουμε, νομίζω θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή μας, περισσότερες πληροφορίες το Σεπτέμβρη πολιτικές αρμοδιοτήτων, αθέμητες πολιτικές, θέματα ενίσχυσης της ε, θέσης των γεωργών στην διατροφική αλυσίδα, με εμπορικές πρακτικές, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω θα τα εξετάσουμε με τη δέουσα προσοχή. Η πολιτική επίσης ανταγωνισμού νομίζω είναι από τα κυριότερα θέματα όσον αφορά την ενίσχυση της ε, θέσης των ε, γεωργών στην ε, διαδροφική αλυσίδα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κοινέ αντιλήψεις, κοινέ ε, απόψεις και συγκλήσεις. Και αυτό θα πρέπει να το αναπτύξουμε μαζί με τις αγορές. Και μιας και μιλάμε για τους ε, για τις αγορές και τους νέους γεωργούς, νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει για την Ένωση. Δηλαδή θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των ε, περιοχών τη υπαίθρου και όταν να βάλουμε υπόψη μα όταν εξετάζουμε του ε, νέου, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανισότητες στι ε, δομές. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι είναι άνω των 65 και είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί ο αριθμό των άνω των 65 στη Γεωργία στο μέλλον. Αν σκεφτούμε λοιπόν την σημασία της ΚΑΠ και, την, ε, και τη στήριξη των νέων γεωργών, ε, θα δούμε ότι αυτά τα μέτρα στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντικά, οπότε θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε ήδη για τα διάφορα κενά στην ε, γεωργική πολιτική και νομίζω ότι θα πρέπει να εποφελθούμε και από τις δημοσίες που είχαμε πρόσφατα τον Ιούνιο για αυτά τα θέματα. Τώρα, να πω και δύο λόγια για τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου Ζούμε σε μια κατάσταση όπου σήμερα πια φαίνεται ο κόσμος να έχει μετατοπιστεί προς όλο και περισσότερο προς μορφές προστατευτισμού. Οπότε πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει η Ευρώπη ότι οι κανόνες ελευθέρου εμπορίου παραμένουν σε ισχύ και ότι αυτό θα πρέπει να ισχύει παγκοσμίω ώστε να ασφαλίσουμε την παγκόσμια ανάπτυξη. Είναι λοιπόν σημαντικό να αφήσουμε τις ε, πολιτικές ελευθέρου εμπορίου ανοιχτές όπως κάναμε μέχρι τώρα και αν κάνουμε νέες συμφωνίες θα πρέπει να τις κάνουμε τηρώντας τις αρχές της ισορροπίας και της ισοτιμίας και σε σχέση με τον γεωργικό τομέα. Το κυριότερο μήνυμα που έχουμε, αλλά και η κυριότερη προϋπόθεση όσον αφορά τα φυτογενομικά είναι το εξής. Τα μέτρα τα φυτογενομικά θα πρέπει να λαμβάνονται για να προστατεύονται για να προστατεύουν την υγεία των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων, θα πρέπει γι' αυτό ακριβώς το λόγο να ανοίξουμε και διάφορες αγορές στους παραγωγούς μας. Αυτό είναι μια αρχή που ανέκαθεν σεβόταν η Ευρώπη. Και μιας και αυτό είναι μια αρχή που σεβόμαστε, θα επιθυμούσαμε βέβαια και οι εταίροι μας να κάνουν το αντίστοιχο. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με την Συμφωνία Θερμορίου με την Ιαπωνία. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να χαιρετήσω τι προόδου που έχει κάνει η Κομισιόν. Αυτό βοηθάει την Προεδρία μα γιατί νομίζω αυτή η συμφωνία ανοίγει νέου ορίζοντες για την Ευρώπη. Και βεβαίω θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό κείμενο συμφωνία αυτή, ελπίζοντα ότι αυτό το κείμενο συμφωνία θα μα δίνει κάποιε θετικέ απαντήσει σε ζητήματα τα οποία παραμένουν άλυτα προ το παρόν όπως επαναδιοργάνωση, το SPS, γεωγραφικές ενδείξεις και άλλες, ε, και άλλες λεπτομερίες και άλλα στοιχεία που εντάσσονται σε αυτή τη συμφωνία. Για τη Μερκοσούρ δεν πω το εξή. Πιστεύουμε ότι για τη Μερκοσούρ θα, μας, θα συνάψουμε συμφωνία ελευθερου εμπορίου με την Μερκοσούρ και σε αντίθεση με την Ιαπωνία είναι μεγάλος εξαγωγέας. Νομίζω πάνω από το 5% των εξαγών του Μερκοσούρ αποτελείται από γεωργικά προϊόντα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι εδώ εμεί αυτό το θέμα βρισκόμαστε σε θέση άμυνα. Οπότε, κατά τη διάρκεια η δικασια σύναψη αυτης της συμφωνιας η γεωργία μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στι συνομιλίε. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να διασφαλίσουμε ως Ευρώπη ότι όλοι οι ευαίσθητοι τομείς μας θα είναι αντικείμενο ε, της δέουσας μεταχείρισης. Τώρα για την Ρωσία και το εμπάργκο, το οποίο υπάρχει από το 2014 και βεβαίως έχει επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό εμπόριο. Υπάρχουν αρκετές ε, χώρες των οποίων η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ακόμα και το 2017, αλλά το 2016 τουλάχιστον οι εξαγωγές όσον αφορά τα τρόφιμα από την Ένωση βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο που είχε ποτέ. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστούν οι προσπαθήσεις ώστε να αναζητήσουμε εναλλακτικέ αγορές. Και νομίζω ότι ό,τι προσπάθειες κάνουμε μέχρι τώρα για την αναζήτηση αυτών των εναλλακτικών αγορών ήταν αποτελεσματικές. Αγορές οι αγορέ γεωργικών προϊόντων είναι πιο σταθεί από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό έχουμε και ανεβοκατεβάσματα στις τιμές. Αυτό βέβαια αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει υποπτία της κατάστασης ε, των αγορών συνεχώς ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της κατάστασης για τους Ευρωπαίους γεωργούς. Από την άλλη μεριά βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γενικότερη κατάσταση όσον αφορά τις γεωργικές αγορές έχει βελτιωθεί και οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί. Πάντως θεωρώ ότι στον ε, τομέα της βιολογικής γεωργίας θα ήθελα να χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για επίτευξη πρόοδου και ελπίζω να είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τις χώρες όπως πρέπει ακριβώς στα πλαίσια του μέρους ε, διαλόγου. Και Πρέπει να σας πω επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των ε, γερικών εδαφών. Αυτό πρέπει να είναι μια από τις προτεραιότητές μας. Η προστασία λοιπόν των ε, γερικών εδαφών σημαίνει θα πρέπει να έχουμε τρόφιμα υψηλής ε, ποιότητας και να υπάρχει η σωστή δυνατότητα παραγωγή του. Γι' αυτό ακριβώ στην Ειδική Επιτροπή Γεωργία θα συζητήσουμε το θέμα των εδαφών ευρέως, όπως ακριβώς και στα πλαίσια του Συμβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι η συγκέντρωση γεών σε κάποια μέρη της Ένωσης είναι ένα θέμα σημαντικό και το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης γεών ίσως να οδηγήσει στην αποχώρηση πληθυσμού από κάποιες περιοχές και αυτό επίσης θα μπορούσε να αποτρέψει και άλλους από το να επιστρέψουν σε αυτές τις περιοχές. Ίσως να έχουμε μάλιστα και απώλειες θέσεων εργασίας, έλλειψη πρόσβαση σε υπηρεσίες και ο αριθμός των θέσεων εργασίας σε αυτές τις περιοχές μπορεί να μειωθεί. Είναι όμως ταυτόχρονα σημαντικό να τηρήσουμε και να σεβαστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης και να μην περιορίσουμε το ελεύθερο εμπόριο εντός της Ένωσης. Ελπίζω πάντως ότι θα είμαστε σε θέση να βρούμε κάποια λύση που θα είναι αποδεκτή από όλους μας. Τώρα. Για τις λοιμώδεις ζωνόσους που έχουν και οικονομικό αλλά και κοινωνικό αντίκτυπο. Νομίζω ότι και η Κομισιόν αλλά και οι χώρες μέλη τακτικά αξιολογούν την κατάσταση σε σχέση με αυτές τις ε, λιμωδείς ε, ζωονόσους, συντονίζουν τις στρατηγικές τους και προσπαθούν να βρουν μια κοινή μεθόδο καταπολέμησης. Στην Εστονία είχαμε πανόλη των και τον τομέα της ε, κτηνοτροφία χείρων επίση αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα και έντονα αυτές τι ασθένειες κι εμεί. Και διάφορα ζώα είχαν μολυνθεί, υποχωρεί ο αριθμό του τώρα, αλλά είχαμε σοβαρέ δυσκολίε στην καταπολέμηση αυτών των ε, φαινομένων με αυτέ τι λοιμώδει ζωνόσου και δεν ξέρω ακόμα αν έχει τελειώσει διαδικασία καταπολέμησης αυτών φαινομένων. Και η γρήπη των πτηνών είχε συζητηθεί και ο αντίκτυπος των μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν για την καταπολέμηση της γρήπης των πτηνών επειδή αυτό το θέμα πραγματικά έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πτηνά ή στα πουλερικά ελευθερά ε, βοσκής επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό το θέμα είμαστε σε θέση να κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη ώστε να εντοπίσουν το ζήτημα και να το καταπολεμήσουν σε συνεργασία πάντοτε με την Κομισιόν. Παρομοίως με το Κοινοβούλιο αλλά και με την Κομισιόν θεωρεί το Συμβούλιο ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το θέμα της μικροβιακής αντοχής, ένα από τα πιο καυτά σημερινά ζητήματα. Εδώ θα πρέπει στην καταπολέμηση να εμπλέξουμε βεβαίω και εμπειρογνώμονες. Και καλωσορίζουμε το νέο σχέδιο δράσης, το οποίο αποβλέπει ακριβώς στην καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Το έγγραφο που θα προκύψει για στρατηγική μας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την καταπολέμηση τη μικροβιακής αντοχή τα επόμενα δύο χρόνια και θα διαμορφώσει τι επιμέρους πολιτικές μας. Τώρα για τις ε, φαρμακούχέ ε, ζωοτροφέ. Σημαντικό αυτό το θέμα όχι μόνο για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για την παραγωγή φαρμακούχων ζωοτροφών στην Ένωση. Αφορά βεβαίως ε, και άλλους τομείς για το τομέα των ε, ζώων συντροφιά και το κυνήγι. Ελπίζουμε πάντοτε να μας στηρίξετε στις προσπάθειες μας ώστε να ολοκληρώσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις και συζητήσεις στο Συμβούλιο. Για τις φαρμακούχες σε αντίθεση με τα κτηνιατρικά φάρμακα. Έχει γίνει προπαρασκευαστική εργασία, αλλά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για τα κτηνιατρικά φάρμακα. Επειδή αυτό ακριβώς σχετίζεται και με τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Και θεωρούμε ότι η φάκελοι αυτή είναι πολύ σημαντική και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι και οι δύο προτάσεις θα προηθούν με συνεκτικό και σαφή τρόπο. Ως Προεδρία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα ώστε να πετύχουμε το, την εντολή, να έχουμε την εντολή διαπραγμάτευση μέχρι το τέλος της θητείας μας. Είναι λοιπόν σημαντικό να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να κατανοήσουμε ότι αν τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιηθούν με τρόπο πιο βιώσιμο, αυτό σημαίνει ότι και χώρες μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά σχέδια δράσης τους για να διευκολύνουν ακριβώς την εφαρμογή της αντίστοιχης οδηγίας. Ο στόχος αυτών των εθνικών σχεδίων δράσης είναι ακριβώς να μειωθούν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, κάτι το οποίο βεβαίως πάντοτε επιφέρει χρήση των φυτοφαρμάκων. Αυτά λοιπόν τα σχέδια δράσης πάντοτε ε, περιλαμβάνουν και εναλλακτικέ λύσεις για την προστασία της ε, υγεία των φυτών και τον περιορισμό των επιπλαβών ουσιών. Αυτά θα είχα να πω ω σύντομη απάντηση στα ερωτήματά σας. Αλλά συνοψίζοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλε αυτέ τις ενδιαφέρουσε ερωτήσει που με υποβάλλατε και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σας καλώ να έρθετε σε επαφή με, τις, με την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου, οι οποίοι μπορούν να σας παράσχουν περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Ήταν χαρά μου που ήρθα εδώ να μιλήσω μπροστά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι καταφέρατε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Όχι πολύ σύντομα, αλλά σίγουρα με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Παρακαλώ τις συμπληρωματικές ερωτήσεις ε, στείλτε τις γραπτός στο Υπουργείο. Θα απαντήσουν οι συνεργάτες ε, όπως μας υποσχέθηκε ο Υπουργός. Πάντως ε, μας περιμένει μια πολύ ενδιαφέρουσα προεδρία εντατικές εργασίες, δύσκολη προεδρία και σύντομη επιπλέον γιατί μεσολαβούν και οι θερινές διακοπές και γύρω στις 15 Δεκεμβρίου σχεδόν ολοκληρώνονται οι εργασίες γιατί έχουμε και τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μετά. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι πάντως, καλές διακοπές, αν και φαντάζομαι ότι οι δικές σας διακοπές θα είναι μάλλον ε, συντομευμένες και περιορισμένες. Πάντως ε, ελπίζω να ξεκουραστείτε κάπως και να αξιοποιήσετε τις διακοπές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε μαζί σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία για την Προεδρία σας και για την Επιτροπή μας, ώστε να έχουμε βελτιώσεις προς το συμφέρον των γεωργών μας πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αρκετά φορτωμένη ημερή διάταξη, όπως είπα και προηγουμένως. Γι' αυτό και ο χρόνος αγόρευσης ε, δεν μπορεί να είναι απεριόριστος. Περνάμε στο επόμενο σημείο, την παρουσίαση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω την κυρία Χέλη Πιχλαγιάμα, που είναι Διευθύντρια για θέματα δικαίου ευρυστεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας που εδρεύει στο Μόναχο. Μάλιστα, ο συνάδελφος Γιάνν με ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσκαλέσουμε, είπα το αξιωματούχο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων ε, με βάση για το θέμα της νομικής προστασίας των βιο... βιοτεχνολογικών εφευρέσεων, κυρίως στη σχέση μεταξύ διπλωμάτων ευρυστεχνίας και δικαιωμάτων βελτιωτών φυτικών ποικιλιών. Επαριλημμένο συζητήσαμε για το θέμα της νομικής προστασίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων και μάλιστα εγκρίναμε ψήφισμα για τα δικαιώματα των ε, βελτιωτών ε, ποικιλιών φυτικών και τα διπλώματα ευρυστεχνίας το Δεκέμβριο του 2015. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών ε, έλαβε υπόψη την, το κατά πόσο μπορούν να κοτοχυρωθούν με δίπλωμα φρυστεχνίας προϊόντα που προέρχονται από κυρίως με βιολογικές μεθόδους. Ε, αυτό το συζητήσαμε επανειλημμένως γιατί ήταν πολύ αφιλεγόμενες οι αποφάσεις ε, του σχετικού Ανώτατου Συμβουλίου Προσφυγών. Στο μεταξύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα ε, σημείωμα διευκρινίζοντας κάποια άρθρα της Οδηγίας 9844 για την προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Η κυρία Πιχλαγιάμα πρώτα θα μας κάνει την παρουσίαση από το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε θερμά και χαιρόμαστε για την ευκαιρία συζήτησης αυτού του τόσο δύσκολου αλλά ενδιαφέροντο θέματος. Παρακαλώ, 10 λεπτά σας αρκούν, άντε 15 το πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σεκέρσκι και ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ε, για να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα σήμερα. Το θέμα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και μας ε, ενδιαφέρει ιδιαίτερος γιατί ε, πριν από 11 μέρες ε, ελήφθη σχετική απόφαση από το Συμβούλιο Προσφυγών. Πολύ σημαντική με σημαντικές συνέπειες. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερη η Επιτροπή σας, η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον για τη δυνατότητα κατοχύρωσης με διπλώματα ευρυστεχνίας ε, εφευρέσεων που αφορούν φυτά τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό θα σας κάνω μια σύντομη επισκόπηση του νομικού πλαισίου αφενός και μετά θα σας παρουσιάσω τις εξελίξεις και τα μελλοντικά βήματα της διαδικασίας αυτής. Στην σύντομη μου εισαγωγή θα επικεντρωθώ μόνο στις ε, εφευρε που αφορούν τα φυτά που είναι το 8% των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Δεν θα επεκταθώ λοιπόν στο σύνολο των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων παρά μόνο σε αυτές που αφορούν τις φυτικές ε, ποικιλίε. Επίσης δεν θα μιλήσω για την προστασία των φυτικών ποικιλιών γιατί αυτό το θέμα της προστασίας των φυτικών ε, ποικιλιών είναι αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και όχι του δικού μας ε, Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η οργάνωσή μας, το Ευρωπαϊκό ε, Γραφείο, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Ευρω... Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ιδρύθηκε το 1973 και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση στη Ευρώπη. Και μάλιστα βλέπετε ότι τα μέλη μας είναι 38 χώρες. Κάτι που σημαίνει ότι το γραφείο μας καλύπτει περίπου 600, 650 εκατομμύρια κατοίκους, πολίτες. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας ε, είναι πολύ ε, κεντρικός παίκτης και παράγοντας στη συνεργασία με άλλα παγκόσμια και διεθνή γραφεία διπλωμάτων ευρυστεχνίας, ε, ιδιαίτερα στο θέμα των διπλωμάτων ευαισθητεχνίας για βιοτεχνολογικά προϊόντα. Εκεί το γραφείο μας, ε, το ΕΠΟ, είναι η φωνή των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευαισθητεχνίας. Και όταν συζητούμε με τα κράτη-μέλη μας, που είναι 38, διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες αιτήσει για βιοτεχνολογικά προϊόντα προέρχονται από το δικό μας το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνία. Δεν, είναι, δεν έχουμε πολλά πολλέ εθνικέ αιτήσει από εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Έχουμε επίση 4.300 επιθεωρητέ που εξετάζουν τι αιτήσει και 7.000 μέλη προσωπικό. Επίσης έχουμε επιστοποίηση ISO και πραγματικά προσβλέπουμε και εφαρμόζουμε πολύ ποιοτικέ διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το νομικό πλαίσιο, τη δυνατότητα κατοχήρωσης, δηλαδή με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Ε, βασικό νομικό πλαίσιο είναι η Σύμβαση του 1973, όπως αναθεωρήθηκε το 2000, η Σύμβαση για τα Διπλωμάτα Ευρεσιτεχνίας του Μονάχου. Επίσης έχουμε και την Οδηγία, 98, την οδηγία του 1998, την Οδηγία Περιθμό 44 του 1998, για την ε, δυνατότητα κατοχύρωσης και περιλήφθηκε η οδηγία αυτή ήδη από το 1999 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και προσθέτει ένα επιπλέον μέσο ερμηνείας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τη Σύμβαση του Μονάχου. Σε ό,τι αφορά την νομολογία του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΠΟ, αυτή η νομολογία είναι πολύ σημαντική εδώ, γιατί για την έτσι και εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων της ε, σχετικής σύμβασης, ε, το Συμβούλιο μας, το Συμβούλιο Προσφυγών και ιδιαίτερα το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών έχει τον τελικό λόγο ε, όταν αποφαίνεται. Και μάλιστα όταν συμπεριλάβαμε και την οδηγία στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, ε, το προβλέπετε το Συμβούλιο Προσφυγών μας δεν μπορεί να παραπέμψει για προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ. Πάντως αναφέρεται σε πολλές αποφάσεις ότι οποιαδήποτε απόφαση για την εφαρμογή την, της σχετικής οδηγίας που γίνεται από το ΔΕΚ είναι πιστικές και λαμβάνονται υπόψη και από το ΕΠΟ και το Συμβούλιο Προσφυγών του ΕΠΟ. Οπότε υπάρχει μια σύνδεση των ομολογιών των δύο δικαιοδοτικών οργάνων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα καταχείριση με διπλώματα ευρυστεχνία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων και κυρίω αυτό που αφορούν φυτά, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι τα συνήθεια κριτήρια κατοχύρωσης ισχύουν εδώ και είναι πολύ σημαντικά. Οπότε, οι βασικέ αρχέ τη κατοχύρωσης, της δυνατότητας κατοχύρωσης είναι ότι η εφεύρεση θα πρέπει να είναι νέα, να περιλαμβάνει μια εφευρετική δραστηριότητα και να είναι επιδεκτική βιομηχανική εφαρμογή. Και όταν μιλούμε για τις καινοτομίε για του νεοτερισμούς, το στοιχείο του νέου, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι κάτι που, ε, που εφευρέθηκε πριν από πολλά χρόνια κάπου, δεν είναι πια καινούριο. Γι' αυτό και το ΕΠΟ, το γραφείο μας, ε, έχει περιλάβει, έχει περιλάβει στη βάση δεδομένων, της, ε, βάση δεδομένων του όλες τι γνώσεις για τα παραδοσιακά φυτά και την κληρονομιά τη και κληρονομιά από πολλά μέρη του κόσμου. Επίσης υπάρχουν κάποια κριτήρια που ισχύουν για τον αποκλεισμό κάποιων εφευρέσεων από τη δυνατότητα κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Τα κριτήρια αυτά εν μέρη εφαρμόζονται και στις βιοτεχνολογικές ε, εφευρέσεις και ιδιαίτερα στη γεωργία. Ο αποκλεισμό εξαιρέσει από την κατοχήρωση περιλαμβάνει εφευρεσει που αντίκυνται στην δημόσια τάξη τα χρηστά ήθη και κάποιες εξαιρεσει αφορούν κάποιες κυριω βιολογικές διαδικασίες για την παραγωγή φυτών ή ζώων. Βέβαια αυτό δεν ισχύει στις μικροβιολογικές ή άλλες τεχνολογικές μεθόδους. Οι διατάξεις αυτές που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα διπλώματα περιστεχνής και τη σχετική οδηγία, την οδηγία 44, οι διατάξεις είναι ταυτόσιμες στι δύο, στις δύο νομοθετικές πράξεις. Επίσης αποκλείονται οι φυτικέ ποικιλίε ή οι φυλέ ζωών που δεν ε, επιδέχονται κατοχήρωση με δίπλωμα με βάση το άρθρο 2 της, Ευ... της ε, οδηγίας ή την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Γιατί για τα θέματα αυτά ισχύει γενική προστασία για τις φυτικές ποικιλίε. Βέβαια, φυτά και ζώα επιδέχονται κατοχύρωση με δίπλωμα ευρυστεχνία εφόσον η τεχνολογική εφαρμοσιμότητα δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο φυτό ή σε μια συγκεκριμένη ζωική φυλή. Σε ό,τι αφορά το βιολογικό υλικό, εφόσον έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον ή παράγεται με τρόπου ή τεχνολογικέ μεθόδου που μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα, ε, γίνεται να κατοχυρωθεί και αυτό. Οπότε, φυτικές ποικιλίε και ζώων γενικώ εξαιρούνται, αλλά φυτά και ζώα μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα υπό όρους και υπό κριτήρια. Οι ε, κυρίως πάντως βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή ζώων και φυτών δεν επιδέχονται κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτέχνικας. Αυτές οι διατάξεις λοιπόν διευκρινίστηκαν και από το Ανώτατο Συμβούλιο ε, προσφυγών του γραφείου μας ήδη από το 1998. Το 1999 είχαμε απόφαση που απέκλει τις φυτικές ποικιλίε από την κατοχήρωση. Με βάση το άρθρο 2 της Οδηγίας για τη Βιοτεχνολογία ε, που προβλέπει ότι φυτά είναι ε, επιδεκτικά κατοχήρωσης, αλλά όχι φυτικές ποικιλίε, αλλά κάποιες τεχνολογικές μέθοδοι, τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Τώρα έχουμε την άλλη απόφαση που αφορά τις κυρίως βιολογικές διαδικασίες ή βιολογικές μεθόδους για την παραγωγή φυτών. Θα ακούσατε ή θα διαβάσετε στις εφημερίδες την απόφαση για την ντομάτα και τα μπρόκολα. Η ερώτηση λοιπόν ήταν αν έχουμε ένα τεχνολογικό βήμα σε μια φυσική, φυσιολογική διαδικασία διασταύρωσης και επιλογής στην, στην βελτίωση η βιολογική αυτή μέθοδος θεωρείται κυρίως βιολογική διαδικασία ή τεχνολογική. Το δικό μας Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών απεφάνθη ότι τέτοιο είδους τεχνολογικό βήμα που συνδυάζει τις φυσιολογικές διαδικασίες διασταύρωσης και επιλογής δεν καθιστά τη διαδικασία από μόνη της τεχνική. Οπότε ανέκυψε το ερώτημα. Αν τα φυτά επιδέχονται κατοχύρωση. Ενώ η συμβατική διαδικασία βελτίωσης δεν είναι ε, κατοχυρώσιμη. Όταν έχουμε ένα φυτό δεν μπορούμε να δούμε από το φυτό πώς έχει παραχθεί, αν έχει παραχθεί δηλαδή με βάση τεχνικές μεθόδους, με μια νέα ε, βελτιωτική τεχνική ή αν παρήχθη από μια συμβατική διαδικασία βελτίωσης, από διασταύρωση δηλαδή ή επιλογή, που είναι κυρίω βιολογική διαδικασία. Τι γίνεται με τέτοιου είδου φυτικά προϊόντα. Επιδέχονται κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνία ή όχι. Ούτε υπάρχουν ξεκάθαρε διατάξει στην οδηγία για τη βιοτεχνολογία, αλλά ούτε και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία υπάρχει σαφή διάταξη που να καλύπτει αυτό το θέμα. Η ανάλυση και αξιολόγηση του θέματο από το Ανώτατο Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου έλαβε υπόψη την οδηγία για τη βιοτεχνολογία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τέτοιου είδου ε, προϊόντα φυτών επιδέχονται κατοχύρωση με δίπλωμα. Οπότε η εξαίρεση ε, για τα φυτά δεν αφορά φυτικά προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε εκ του σύνεγγης το προπαρασκευαστικό υλικό της ε, οδηγίας για τη βιοτεχνολογία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να αποκλείσει και τα φυτικά προϊόντα που παράγονται από κυρίως βιολογικές διαδικασίες που εξαιρούνται της ε, κατοχυρωσιμότητας. Και μάλιστα αυτό προβλέπει το, το σχετικό μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έκτοτε έχουμε ε, διακόψει όλες τις διαδικασίες εξέτασης της κατοχύρωσης ή ανακοπής σε περίπτωση που είχαμε φυτικό προϊόν που ε, παρήχθη από κυρίως βιολογική διαδικασία. Γιατί όταν ε, υπάρχει αφιβολία για την εφαρμογή μιας νομικής διάταξης, είμαστε υποχρεωμένοι να ε, διακόψουμε τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να μην βλάψουμε κανέναν ενδιαφερόμενο. Τα κράτη-μέλη κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού ε, δεν, κατέληξα, δεν σε συμπέρασμα. Εμεί υποβάλαμε μία τροποποίηση του εφαρμοστικού κανονισμού και με βάση την πρόταση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστεχνία στις 29 Ιουνίου αποφάσισε να τροποποιήσει το, τα σχετικά άρθρα 27 και 28 του, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Διπλώματα Ευρυστεχνίας, ώστε ζώα ή φυτά που παράγονται αποκλειστικά από κυρίω βιολογικέ μεθόδου, εξαιρούνται τι δυνατότητε κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Και αυτή η αλλαγή τη νομοθετική διάταξη ισχύει για όλε τι διαδικασίε που ήδη εκκρεμούν, για όλε τι αιτήσει που εκρεμούν μέχρι που εκκρεμούν την 1η Ιουλίου του 2017 όταν, όταν έληφθη η απόφαση και ισχύει όχι μόνο για τις εκκρεμίες, αλλά και για τις μελλοντικέ αιτήσει για διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτό που κάνει τώρα το γραφείο μας είναι ότι όλες οι διαδικασίες και εξέτασης και ανακοπής θα συνεχιστούν σταδιακά, με βάση όμως τους νέους κανόνες. Οπότε, ένα προϊόν φυτού που είναι αποτέλεσμα κυρίως βιολογικής διαδικασίας εξαιρείται από την κατοχήρωση. Οπότε σε τέτοια περίπτωση η αίτηση θα απορρίπτεται για δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Οι κατευθυντήριε γραμμέ για την ε, εξέταση που είναι, ισχύουν για του επιθεωρητέ ε, περιλαμβάνουν και κάποιε πληροφορίε και για το κοινό και θα τροποποιηθούν ανάλογα με τη τελευταία απόφαση. Οι κατευθυντήριε γραμμέ θα δημοσιευθούν τον Οκτώβριο και θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο του τρέχοντο έτου. Ταυτόχρονα και ήδη από το 2016 έχουμε στενή συνεργασία με το Κοινοτικό Γραφείο ε, Φυτικών Ποικιλιών, το CPVO, ώστε να ε, εξοικειωθούμε ημέν με τα συστήματα και τις διαδικασίες των ΔΕ και να αξιοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων μας και το υλικό που έχουμε, τις πληροφορίες που έχουμε για να αποφύγουμε προβλήματα ή να, να μην αγνοούμε πράγματα σημαντικά. Επίσης από κοινού με το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών θα ενημερώνουμε το κοινό για τις ε, εργασίες μας σε μια δημόσια διάσκεψη που θα γίνει τον Νοέμβριο φέτος στις Βρυξέλλες. Μια κοινή διάσκεψη των γραφείων του διπλώματος, δηλαδή του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνής και του Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά μέτρα, για τις αιτήσει διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για τα φυτά. Έχουμε κάποιες ευαίσθητες περιπτώσεις και μια σχετική ομάδα για τις ευαίσθητες περιπτώσεις, για τις ευαίσθητες υποθέσεις. Εκεί εξετάζουμε εκ του σύνεγγυ όλες τις αιτήσει ε, για διπλώματα που αφορούν φυτά ή φυτικά προϊόντα. Και εκεί έχουμε την συνδρομή δικηγόρων Οπότε οι επιθεωρητές μας και οι υπηρεσίες μας λαμβάνουν υπόψη και τις κοινωνιολογικές αλλά και τις ηθικές πτυχές κατά την εφαρμογή των εξαιρέσεων από τη δυνατότητα κατοχήρωση με δίπλωμα ευρυστεχνίας. Επίσης υπάρχει εθνικό ενδιαφέρον για τις πρακτικές και τις εργασίες μας. Μέχρι στιγμής πάντως υπάρχει συνεννόηση ως προς τα αποτελέσματα και κοινή αντίληψη παρά κάποιες διαφορές απόψεων. Και φυσικά ζωηρό ε, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και το ευρύ κοινό για τις εργασίες του γραφείου μας. Αυτά εν εισαγωγή και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε απορίες σας και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με ναι, πρώτο τον κύριο Χαΐτεμα που έχει την πρωτοβουλία αυτή τη συνάντηση. Παρακαλώ. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Διευθύντρια για την παρουσία της εδώ, καθώς και για την παρουσίαση του θέματος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που βλέπω ότι το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών δέχεται τις συμβουλές και συστάσεις του Κοινοβουλίου Ήδη από το 2015 μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή Γεωργίας και ταχθεί υπέρ της προστασίας της δυνατότητας ναι, ε, της δυνατότητας προστασίας της φυτικών ειδών. Έχω τρεις πιο λεπτομερείς ερωτήσεις που θα ήθελα να σας υποβάλω. Πρώτα, για την ώρα Υπάρχουν εκατοντάδες αιτήσει για ευρεσιτεχνική προστασία για φυτά που προέρχονται ιδίως από ουσιοδός βιολογικές διαδικασίες. Τώρα όμως το ΕΠΟ έχει ε, αποφασίσει να τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταλλαξιογέννηση πρόκειται να τη λάβει υπόψη του για την ε, προστασία το ε, Γραφείο εστεχνιών Και τρίτο, προϊόντα τα οποία βασίζονται σε ουσιοδός βιολογικές διαδικασίες θα παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογή οποιονδήποτε ε, ευρεσιτεχνιών ακόμα και αν υπησέρχονται σε αυτά και κάποιες ε, τεχνικές διαδικασίες βελτίωσης ανεξάρτητα από την απόφαση που ελήφθη από το Γραφείο Τεχνιών στις 29 έκτου. Έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε μετά. Παρακαλώ κυρία Schreier, που επίσης είναι Ολλανδέζα. Ευχαριστώ να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας. Το ΕΡΚ είχε δουλέψει πάνω σε ένα ψήφισμα για αυτό το θέμα το 2015 και η ίδια η χώρα μου, οι κάτω χώρες, ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή του 35% στις παγκόσμιες αγορές αυτών των σπόρων. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική που ανοίγει το δρόμο για διάφορες ποικίλε φυτών. Όμως θα ήθελα να μάθω τι συμβαίνει όταν ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί. Θα πρέπει να πάνε στα δικαστήρια οι κάτοχοί τους για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Ε, τι θα γίνει λοιπόν στον τομέα αυτό. Τι θα γίνει με τις παραδοσιακέ μεθόδου βοηθήσει των φυτών και τι νέε Μετά να ρωτήσω, αυτοί που κάνουν βελτίωση φωτών, φυτών μπορούν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένε ποικιλίε και τι γίνεται, ξαναλέω, με τις ε, παρουσιακέ μεθόδους βελτίωσης σε σχέση με τις νέες αυτές μεθόδους. Η Μονσάντο αλλά και άλλοι ήθελα από ανακοίνωσαν θα προσφύγουν κατά τι αποφάσει αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι επιπτώσει θα έχει αυτό, δηλαδή πώ θα μπορούσαν να παρακάμψουν την ε, απαγόρευσή σα ή να ανατρέψουν ακριβώ την απόφαση. Και πώ θα ε, μπορέσετε να παρακολουθήσετε ακριβώ την εφαρμογή της απόφασης και για την, ε, για την περίοδο αξιολόγησης ένα-δύο έτη για την αγορά σπόρων δεν υπάρχει απαγόρευση παγκόσμια όσον αφορά τις παρουσιακές μορφές βελτίωσης. Μήπως η Μονσάντο και άλλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για να κάνουν τη δικιά τους πολιτική. Πώς θα το αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ. Ο κ. Σταραμπέλα, δύο λεπτά. Κύριε Σταραμπέλα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε ότι το γραφείο σας είναι διακυβερνητικό γραφείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και υπάρχει σοβαρή λήψη ανθρώπινων πόρων. Οπότε εκφράζω την ε, συμπόνια μου προς εσάς, την κατανόησή μου, για αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Γιατί μιλάμε σήμερα. Κάποια φύτα ε, βελτιώνονται με, με φυσιολογικό τρόπο όπως θα ξέρετε. Υπάρχουν βέβαια νέες μέθοδοι όπως η μικρολογική πτωγέννηση, αλλαξιογέννηση, συγγνώμη, Υπάρχουν λοιπόν τρόποι που δυστυχώ δεν μα επιτρέπουν να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ αυτών των τρόπων βελτίωση. Το είπαν και προηγουμένω εξάλλου τα διπλώματα αυτά αφορούν και φυτά ή μεθόδους που είναι πολύ φυσικές. Οπότε η βιομηχανία βράχει πρόθεσμα και μέσω πρόθεσμα θα καλύψει την ε, πλειοψηφία ακριβώς της βιοποικιλότητας και θα προσπαθήσει να την ελέξει μέσω ακριβώς της παραγωγής αυτών των βελτιώσεων. Και αυτό είναι ένας σημαντικός κίνδυνος. Ε, συμφωνείτε λοιπόν ότι ε, μήπως θα έπρεπε ακριβώς να απαγορεύσουμε οποιοδήποτε δίπλωμα όσον αφορά τα φυτά και να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να απλά και μόνο να χρησιμοποιηθούν άλλες ε, μεθοδοί πιο παρουσιακές, πιο φυσικές κατά κάποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Κυρία ε, Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Κατά βάση είμαι απογοητευμένη με αυτά που κάνετε, δηλαδή με την αντίδρασή σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπετε ότι θέλετε να βγάλετε απ' έξω την συμβατική βελτίωση, την οποία όμως ορίζεται πάρα πολύ στενά το πρόβλημα με τις μεταλλακτικές ε, βελτιωτικές τεχνικές, εκεί τα είπατε εσείς δεν θέλω να δώσω περισσότερες ερμηνείες, είπατε όμως ότι και πρέπει από πίσω να υπάρχει μια βιοτεχνολογική επινόηση. Από την άλλη μεριά επιτρέπεται να δίνονται έβρεση τεχνίες για ορισμένα γενετικά χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, ε, εγώ τα βλέπω αυτά πολύ επικριτικά. Εάν εξετάσει κανείς με ποιον τρόπο έχει γίνει, έχει προσθεθεί το χαρακτηριστικό, εάν υπάρχει ήδη στην φύση δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι η αξία της τεχνολογικής επινόησης, δηλαδή απλώς το εντόπισε. Αυτό που κάνετε εσείς είναι να ανοίγετε μια επιχείρηση δισεκατομμυρίων ευρώ σε αξία για την αγροτεχνική ε, οικονομία στο μέλλον δηλαδή θα μπορούν να βελτιώνουν κάποια ε, φυτά, δεν θα γνωρίζετε καν όμως, θα γνωρίζουν μάλλον καν ε, αυτοί που τα προωθούν τα πράγματα αυτά, εάν το χαρακτηριστικό αυτό υπήρχε ήδη. Στην ουσία βγαίνετε και πουλάτε την γενετική κληρονομιά σε επιχειρήσεις. Δεν ξέρω τι θα κάνετε στο μέλλον εν ώψη αυτών των μεγάλων παρατηριών του νόμου, ας το πω έτσι. Υποθέτω ότι θα έχετε πλήθος αιτήσεων στο μέλλον. Τι προβλέπετε ωστόσο. Θα εξετάζετε την επίδραση των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων ενδεχομένως για να βάζετε κάποιο φρένο. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που προβλέπετε. Και άλλη μια ερώτηση για τον καθορισμό των ε, διαδικασιών για τις αποφάσεις έχουν περιληφθεί και ενδιαφερόμενοι. Έχετε ακούσει τις γνώμες των οργανώσεων ε, των ε, γεωργών, των οργανώσεων προστασίας καταναλωτών, μη κρατικών οργανώσεων που θεωρούν ότι η ζωή δεν είναι δυνατό να είναι αντικείμενο ευρεσιτεχνιών. Εσείς τώρα κύριε Άγνιο. Πρώτα ευχαριστώ. Δεν είμαι ο μόνος στην αίθουσα που νομίζει ότι το θέμα περιπλέκθηκε περισσότερο. Και κάπως έμεινα άφωνος με, αυτά, με κάποια από αυτά που είπατε. Είπατε ότι γίνεται να καταθέσουμε ή να λάβουμε τέλο πάντων δίπλωμα για ένα ζώο αλλά κάτι το οποίο υπήρχε ή προπήρχε. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Το ίδιο και για ένα φυτό ή για μια μορφή καλλιέργεια. Είναι κάτι σαν τα ανθρώπινα όντα. Δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίστηκε τώρα. Να μου απαντήσετε. Θεωρούσα κάποια θέματα για το σε κάποια θέματα, για κάποια πράγματα θα πρέπει να υπάρχει δίπλωμα ευρεσιτεχνία, μου φαίνεται κάπω κοντόφθαλμο αυτό. Γιατί όποιο ε, κάνει αυτέ τι ε, έρευνε αναμένει κάποιο κέρδο και κάποια απολαβή. Και βέβαια ε, αυτά τα διπλώματα δεν διαρκούν για πάντα. 20 χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά να μου το επιβεβαιώσετε αν έχετε καλοσύνη. Ευχαριστώ κύριε εγώ θα συμφωνήσω με την πλειοψηφία που θεωρεί κάπως απογοητευτικά τα όσα έχετε, έχετε επιτύχει ως τώρα. Εγώ υπενθυμίζω κάποια ψηφίσματα ήδη από το 2011 με μεγάλη πλειοψηφία και αν εξετάσετε τα πράγματα πιο προσεκτικά θα βρείτε τόσα πολλά παράθυρα στην νομοθεσία τα οποία έχετε διατυπώσει εσείς που θεωρώ ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν πολλά στις πρακτικές που ισχύουν τώρα. Τι γίνεται και με, τις με τα 200 διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία έχετε ήδη απονείμει. Τι θα γίνει στο μέλλον. Μια μετάλλαξη που ενδέχεται να προκύψει τυχαία. Μπορεί και αυτή να πατενταριστεί. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά παράθυρα λοιπόν στις ρυθμίσεις αυτές. Βεβαίω το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών ζει από την απονομή πατεντών. Δεν πιστεύω λοιπόν να εμφανείται πολύ περιοριστική, διότι καταρχήν η δουλειά σας αυτή είναι. Και ε, υποθέτω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει πολύ η πρακτική σας. Τώρα ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Πρόκειται για αυτή την ε, συζήτηση μεταξύ Καρλσπεργκ και Χάινεκεν για ένα είδος ε, Βίνης που ε, έχει υποστεί μια ε, γενετική μετάλλαξη και ε, πού θα καταλήξει εν τέλει, εν τέλει. Αυτό θα μπορούμε τελικώς να πίνουμε την πύρα ήσυχη. Σας ευχαριστώ. Να καλωσορίσω και κάποιους καλεσμένους μας, επισκέπτες που θα καταληξει εν τελει αυτο θα μπορουμε τελικως να πινουμε την πυρα από τον κύριο Χαϊτέμα Καλώ ήρθατε. Παρακολουθείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη συζήτηση. Και ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα αυτό που πραγματευόμαστε. Ο κύριο Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω κύριε Διευθυντριά που ήρθατε στην Επιτροπή μα, Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή για να παρακολουθήσω όλη σα την παρουσίαση και μάλιστα μερικά σημεία επαναλαμβάνουν τους τα σχόλια των προλαλισσάντων. Εγώ θα σταθώ κυρίως στο θέμα της καινοτομίας, της ευρηματικότητας. Ε, ε, αυτό είναι χαρακτηριστικό κριτήριο που απαιτείται, η εφευρετικότητα. Επίσης, τι γίνεται με την προστασία. Τι γίνεται σε περίπτωση που ο κλάδος ε, οικειοποιηθεί ένα γενετικό πόρο που σήμερα ανήκει στο δημόσιο. Τι θα συμβεί, τι προστασία επιτρέπεται. Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος Ταραμπέλα, το θέμα είναι τεράστιο και ιδιαίτερα περίπλοκο και το διακύβευμα τεράστιο. Μιλήσαμε για κάποια μεγαθύρια πολυεθνικές ε, Συνζέντα με μια Κινέζικη, Μονσάντο με την Μπάγερ, ε, ίσως το γραφείο θα έπρεπε να ενισχυθεί με πόρους και δυναμικό. Γιατί πώς θα ε, διενεργήσει διεξοδικούς ελέγχους, κάτι που απαιτείται για τη χορήγηση ε, διπλωμάτων ευρυστεχνίας. Δεν μπορεί με λίγα μέσα να ανταποκριθεί στο έργο του. Επίσης, το θέμα της φυτικής ποικιλία. Και αυτό είναι περίπλοκο ζήτημα και κατά τη γνώμη μου ε, αυτό είναι το ζήτημα που βρίσκεται και στο επίκεντρο της συζήτησης. Και έτσι αυτό το κενό εκμεταλλεύονται οι πολυεθνικές και προσπαθούν να οικειοποιηθούν τέτοιο γενετικό υλικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Θα καταλάβατε πόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κατά της δυνατότητας κατοχύρωσης της ζωής με δίπλωμα ευαισθητεχνίας. Είναι ανεπίτρεπτο κάτι τέτοιο. Επίσης, τι θα πρέπει να αλλάξει, οι νομοθετικές διατάξεις ή τίποτα άλλο για να αποφευθεί τέτοια δυνατότητα να κατοχυρώνουμε την ίδια τη ζωή με δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Μιλήσαμε για τους σπόρους, πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ε, για τους γεωργούς, η πρόσβαση τους ε, σε σπόρους. Και αν ε, δοθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για σπόρους, μήπως ε, θα διατρέξουν κίνδυνο οι γεωργοί σε ό,τι αφορά την πρόσβασή τους σε, σε σπόρους, γιατί μιλήσαμε για διάφορα είδη φυτών. Θα πρέπει όμως ο κάθε γεωργός να μπορεί να βελτιώνει τους σπόρους του. Θα πρέπει να έχει τέτοια ελευθερία και πρόσβαση σε διάφορες γενετικές επιλογές. Και αν υπερέχει εδώ το, δίπλωμα, το δίκαιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας περιορίζονται οι ελευθερίες των γεωργών. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγκίνες. Πολύ, πολύ τεχνικό το θέμα και από την άποψη των βελτιώσεων, τεχνικά δηλαδή, αλλά και την νομική άποψη. Γι' αυτό και ρωτώ την αφελή ερώτηση. Παρακολούθησα χθε, νομίζω, μια εκπομπή στο BBC, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, σχετικά με την βελτίωση ποικιλιών πορτοκαλιών που είναι πολύ εύκολο να τα ξεφλουδίσει κανεί. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Χρειάζεται 8 με 10 χρόνια για να φτάσουν στο στάδιο όπου θα έχουμε αυτά τα πορτοκάλια που είναι εύκολο να ξεπλουδιστούν. Υποθέτω ότι αυτά προστατεύονται κάποια ευρεσιτεχνία, διότι κάποιο θέλει κέρδο από την επένδυσή του. Ή εν πάση περιπτώσει πώ γίνεται αυτό. Είπε ο Άγνιου πριν ότι οι επιχειρήσει επενδύουν χρήματα και χρόνο για ε, τη χρήση ε, βελτιωτικών τεχνικών εκτός GMO, εκτός δηλαδή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αυτή την ερώτηση κάνω. Τα περισσότερα από τα λουλούδια μας, άλλα φυτά, ε, λαχανικά και ε, φρούτα έχουν χρησιμοποιήσει πολύ προηγμένες τεχνολογίες για να φτάσουν στο στάδιο που βρίσκονται σήμερα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Ε, πόσο ενεργειοβόρα θα είναι αυτά τα τεχνητά πορτοκάλια ή τα ευκολοξεφλούδιστα πορτοκάλια. Η κυρία Κάντεμπαχ. Thank you very much. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την αρχική σας παρέμβαση. Ίσως λοιπόν να έχετε απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Παρ' όλα αυτά να με επιτρέψετε να τις κάνω. Ένας εκπρόσωπος του ΕΠΟ είπε ότι υπάρχουν 320 αιτήσει για φυτά και ζώα που εκκρεμούν. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη των αποφάσεων. Δεύτερη ερώτηση, γιατί ήμουν σκιώδη συζητήτρια για θέματα, για την οδηγία μάλλον αναπαραγωγής φυτών. Ξέρετε ποια ήταν η σαφής θέση του Κοινοβουλίου επ' αυτής. Ερώτηση λοιπόν, Ευρεστιχνίε για φυτά προκαλούν σημαντικά προβλήματα στους βελτιωτέ, διότι δεν υπάρχει το προνόμιο του βελτιωτού. Τι έκανε το ήπιο για να κατανοήσει τι επιπτώσει των αποφάσεών του στον τομέα, στον τομέα των βελτιώσεων. Εσείς κύριε Φλάνναγκάν Πολύ ενδιαφέρουσα και τεχνική η παρουσίασή σας. Διαρωτώ με, έχετε καταχωρήσει ε, ε, αιτήσει ευρεσιτεχνία για την ιατρική κάναβη ή έχετε κάποιες που περιμένουν τη σειρά τους αιτήσει δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, μήπω θα ήθελε το λόγο. Ο κύριος Γκάλ. Αλλά παρακαλώ χρόνου φίδου. Ή μήπως δεν θέλετε καν να μιλήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Πίλα Γιάμα και τους ε, ευρωβουλευτές που έλαβαν το λόγο για αυτό το πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Ε, ε, μετά την απόφαση των ΟΤΑ του Συμβουλίου Προσφυγών του ΕΠΟ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε υπόμνημα για την διευκρίνηση της βούλησης του νομοθέτη για μια οδηγία που έχει ήδη 20 χρόνια ζωής και στόχος δεν ήταν να δοθούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας για προϊόντα που είναι αποτελέσματα κυρίως βιολογικών διαδικασιών. Γι' αυτό και εκδώσαμε το υπόμνημά μας. Και το Συμβούλιο το Φεβρουάριο φέτος ε, εξέδωσε σχετικά συμπεράσματα και επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας τροποποίησε το εφαρμοστικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Πατέντες και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου και βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θίξατε πολλά ζητήματα ενδιαφέροντα και αρκετά περίπλοκα από τεχνική άποψη. Χρειάζεται περαιτέρω εξέταση για να δοθούν απαντήσεις. Πάντως, πρόθεση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να εξετάσει διεξοδικά όλα τα επιμέρους ζητήματα και να συζητήσει με τα κράτη-μέλη ε, για να εξακριβώσει τις λύσεις που έχουν δώσει και σε μεταγενέστερο στάδιο θα σας δώσουμε το αποτέλεσμα όλων αυτού του προβληματισμού. Κυρία Διευθύντρια, ήρθε η ώρα παρακαλώ να δώσετε τις απαντήσεις, αλλά για το πολύ ένα δεκάλεπτο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας για τις ερωτήσεις τους. Αν μου δίνετε ευκαιρία να απαντήσω μόνο σε ένα δεκάλεπτο τι να πω. Θα κάνω ό,τι μπορώ, πάντω θα βάλω τα δυνατά μου. Προσπάθησα να ομαδοποιήσω μερικέ ερωτήσει, θα προσπαθώ ίσω να μιλήσω και γρήγορα για να απαντήσω σε όσο το δυνατό περισσότερε ε, ερωτήσει. Αν κάτι μου διαφύγει, το ξεχάσω να μου το επισημάνετε. Για τα στατιστικά στοιχεία. Μα ρωτήσατε για τι εκκρεμεί αιτήσει και για τι ήδη αποδεκτέ αιτήσει που έχουν. Είχαμε περίπου 300 ε, αιτήσει εκκρεμεί για φυτικά προϊόντα που επηρεάζονται από τις τελευταίες αποφάσεις τώρα και οι διαδικασίες για τη χορήγηση διπλώματος ή για την ανακοπή έχουν, είχαν διακοπή αλλά έχουν ε, σταδιακά επανέλθει στην εξέταση και προσπαθούμε μέσα σε 12 μήνες να διεκπεραιώνουμε την εξέταση των αιτήσεων και τις ανακοπές μέσα σε 15 μήνες. Θα τηρήσουμε αυτό το πρόγραμμα, εκτός και αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία είναι πιο χρονοβόρα. Πάντως, μέσα σε ένα, ενάμιση χρόνο το πολύ, θέλουμε να διεκπαιρεώσουμε όλες τις εκκρεμείς αιτήσει για χορήγηση διπλώματος ή τις ανακοπές, τις αντιρρήσεις. Περίπου 80 διπλώματα δόθηκαν στο παρελθόν πάντως για τέτοιου είδους φυτικά προϊόντα Οπότε αυτά πια δεν εμπίπτουν στην ε, δικαιοδοσία, στην αρμοδιότητα του γραφείου μας. Βέβαια, μία πατέντα έχει ισχύ το πολύ 20 χρόνια. Και όσο είναι ενισχύ, ο δικαιούχος πρέπει να, καταλάβει, να καταβάλει ετησίως ένα τέλος, μια εισφορά, εκεί που έχει εγκριθεί το δίπλωμά του. Αλλιώς ε, ε εκπνέει. Και περίπου 80 τέτοια διπλώματα δόθηκαν ε, με βάση τις στατιστικές μας, όπως σας είπα, και έχουν υποβληθεί στα συμβούλια, αλλά περίπου μισά έχουν χάσει πια την ισχύ τους λόγω μη καταβολής των ε, απαραίτητων τελών. Αν και κάποιοι δικαιούχοι ε, είτε αναλαμβάνουν κάποια δράση είτε αφήνουν το δίπλωμά τους και εκπνέει. Πάντως δεν είναι όλα, επαναλαμβάνω, ακόμη ενισχύ από αυτά τα 80 που χορηγήσαμε. Τώρα, τι γίνεται μετά την λήψη της απόφασης. Ήδη αυτό συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γραφείου και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ε, είπε, όπως και πολλά κρατημέλη, ότι αυτό που θα κάνουμε εμείς στο γραφείο μας είναι ότι κάποια στιγμή σε έναν 1,5 χρόνο όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της δεκπεραίωσης των αιτήσεων θα υποβάλουμε ενημέρωση στα κράτη-μέλη για την κατάσταση και θα συγκεντρώσουμε τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για το τι, ποια ήταν η μοίρα των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί. Επίσης, ρωτήσατε ε, για την ανάμειξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλων ομάδων συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει τη μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή του. Εκεί ε, εκπροσωπούνται πολλές οργανώσεις και μέλη ad hoc που ορίζονται στην Επιτροπή προκειμένου να έχουμε τη, την ενημέρωση και από τους χρήστες. Πάντως δεν βάλαμε υπόψη όλες τις πληροφορίες. Για το συγκεκριμένο θέμα, πολλές οργανώσεις χρηστών έστειλαν επιστολές στο γραφείο μας και σχόλια με προτάσεις και σας υπόσχομαι ότι τέτοιες είδους πρωτοβουλίες δεν παίρνουν απαρατήρητες. Υπάρχουν κάποια θέματα που τα λαμβάνουμε υπόψη και άλλα που φυσικά που δεν τα δεχόμαστε. Γιατί οι χρήστες έχουν διαφορετικά ε, σχόλια και απόψεις, δεν μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη όλα, παρόλο που τα εξετάζουμε όλα. Τώρα έρχομαι στα πιο τεχνικά ζητήματα. Ένα-δύο ερωτήσεις αφορούσαν κάποια θέματα όπως η, ιατρική κάναβης. Δεν έχω πληροφορίες. Επίσης, τα πέτατες για τα χλάδια, peer patent, δεν ακούσαμε καλά, ούτε γι' αυτό έχω πληροφορίες, οπότε δεν μπορώ να σας ε, ενημερώσω ιδιαίτερα αν εκκρεμούν και όλα οι διαδικασίες. Και για την ιατρική χρήση της κάναβης ε, δεν έχω γνώση. Μιλήσατε για την ελευθερία των βελτιωτών και την ελευθερία των γεωργών και κατά πόσο αυτή παρεμποδίζεται από διπλώματα ευρύς που έχουν χορηγηθεί. Θα το ξέρετε κι εσείς, αλλά το επισημαίνω παρόλα αυτά. Υπάρχει μια μία συμφωνία για, την, για το ομοιόμορφο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των κυρώσεων από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω αυτά τα, αυτοί οι μηχανισμοί να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Πάντως, στην Συμφωνία για τη Σύμβαση του Μονάχου προβλέπονται κάποιες εξαιρέσεις για τους βελτιωτές, ιδιαίτερα αν έχουμε ένα νέο δίπλωμα για, τα, για ορισμένα κρατημέλη, για όλα τα κρατημέλη, αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει συμφωνία θέσεως σε ισχύ ή κάποιες δράσεις ε, σε εθνικό επίπεδο, κάτι που ήδη ισχύει σε ορισμένα κρατημέλη, αλλά όχι σε όλα, ώστε να θεσπιστεί η εξαίρεση για τους βελτιωτές ε, στην εθνική νομοθεσία. σε ό,τι αφορά τη μεταλλαξιογένεση και τα εγγενή χαρακτηριστικά. Η μεταλλαξιογένεση, όπως εξηγήσαμε και στο έγγραφο που υποβάλαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο, η τεχνική μεταλλαξιογένεση θεωρείται ως τεχνική διαδικασία. Η τυχαία μεταλλαξιογένεση είναι τυχαία υποθετική και όπως ανέφερε και η κυρία Μαγκίνες, Τα αποτελέσματά της είναι αβέβαια και άγνωστα. Μπορεί να είναι και ανεπιθύμητα, οπότε δεν είναι σταθερό ή δεδομένο το αποτέλεσμα μιας τυχαίας μεταλλαξιογένεσης. Οπότε μια τέτοια μέθοδος είναι πολύ πιο χρονοβόρα. Πάντως οι νέες τεχνικές βελτίωσης που περιλαμβάνουν κάποιες μεταλλάξεις θεωρούνται ως τεχνικές εφευρέσεις, τεχνικές μέθοδοι. Οπότε οι νέες μέθοδοι βελτίωσης δεν θεωρούνται ουσιοδός ή κυρίως βιολογικές διαδικασίες, παρά τεχνικές διαδικασίες. Ε, και μια ερώτηση για τα εγγενή χαρακτηριστικά. Αυτή η ερώτηση όμως είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα. Δεν ξέρω μου επιτρέπετε να επισέλθω σε τόσο τεχνικά θέματα. Το θέμα των εγγενών χαρακτηριστικών και τα διπλώματα για τέτοια εγγενή χαρακτηριστικά. Καταρχήν, τα εγγενή χαρακτηριστικά υπάρχοντος φυτού δηλαδή γνωστού φυτού, με βάση τους νέους κανόνες όπως έχουν διαμορφωθεί, δεν επιδέχονται κατοχύρωση. Για παράδειγμα, θέλω, εγώ θέλω κόκκινα αγκούρια. Δεν μου αρέσουν τα, τα πράσινα, τα ανοιχτά πράσινα. Θέλω κόκκινα αγκούρια. Με βάση τους νέους κανόνες, αν υποβάλω αίτηση διπλώματος για κόκκινα αγκούρια, ε, εμπίπτει αίτηση στην εξαίρεση. Θα μπορούσα όμως να ζητήσω αίτηση, αλλά μου λείπει ο τεχνικός όρος. Το χαρακτηριστικό του κόκκινου χρώματος το αγγούρι αν ε, επιτυχάνεται με τεχνικές μεθόδους, ε, μπορεί να κατοχυρωθεί. Τα φυσικά, φυσιολογικά όμως αγκούρια δεν εμπίπτουν στην προστασία. Αλλά έχουμε και το άρθρο 5 της Οδηγίας για τη Βιοτεχνολογία που επεκτείνει την προστασία και σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, σε εθνικά δικαστήρια μπορεί να προσφύγει ο βελτιωτής και να πρέπει να αποδείξει αν η διαδικασία που χρησιμοποίησε ήταν κυρίως βιολογική ή τεχνική για να επιτύχει το κόκκινο χρώμα. Εκεί χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Θα έπρεπε να σας κάνω τρία τέταρτα τουλάχιστον διάλεξη για το δίκαιο ε, διπλωμάτων ευρυστεχνίας και δεν μου το επιτρέπετε. Γι' αυτό και ομολογώ ότι η απάντησή μου είναι κάπως ασαφής, αλλά ελπίζω στη δημόσια διάσκεψη που θα οργανώσουμε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών να δώσουμε πιο διεξοδικές ε, εξηγήσεις Γι' αυτό και σας προσκαλώ τώρα σε ένα δεκάλεπτο που μου δώσετε, έκανα ό,τι μπορούσα. Ήδη ε, πλησιάζω προς το τέλος τη, του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου, γι' αυτό και δεν προλαβαίνω να σας δώσω πιο λεπτομεριακές εξηγήσεις. Ποιο είναι το συμπέρασμα. Τα εγγενή χαρακτηριστικά επιδέχονται κατοχύρωση, εφόσον απομονώνονται από το φυσικό περιβάλλον τους με βάση τη Οδηγία για τη Βιοτεχνολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Διπλώματα Ευρυστεχνίας. Το θέμα είναι πόσο επεκτείνεται η προστασία και υπό ποιου όρους και τι αποδείξεις, τι τεκμήρια θα πρέπει να ε, καταθέτει ο βελτιωτής για το ότι δεν παραβαίνει τη διαδικασία. Αλλά γι' αυτό θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Πάντως, παραλαμβάνω, είναι σημαντικό να έχουμε το ομοιόμορφο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνία και ελπίζω να διεκπαιρεωθούν οι σχετικέ εργασίε το συντομότερο δυνατό. Μου ζητήθηκαν κάποια παραδείγματα φυτών και ζώων. Κάθε ζώο φυσικό ή κάθε φυτό φυσικό που το βλέπουμε στους αγρούς δεν μπορεί να κατοχυρωθεί από δίπλωμα γιατί δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι γνωστά αυτά τα είδη των φυτών και των ζώων. Αν ναι, όμως έχουμε ένα ζώο στο οποίο έχουν περιληφθεί κάποια, κάποιες ιατρικές, ε, θεραπευτικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, έχουμε μια εφεύρεση ώστε να συμπεριλαμβάνουμε ένα γονίδιο στην Αγελάδα και να έχει το γάλα της θεραπευτικό χαρακτήρα οι κανονικές φυσιολογικές αγελάδες ε, προστατεύονται, δεν καλύπτονται από δίκαιο ευρεσιτεχνία, αλλά η αγελάδα με θεραπευτικό γάλα μπορεί να εμπίπτει σε, τέτοια προστασία, σε τέτοιο δίπλωμα. Και για την ε, κατοχήρωση των ζώων λαμβάνονται και άλλα κριτήρια υπόψη. Ε, τα χρηστά ήθη, για παράδειγμα, η δεοντολογία, το θέμα της μη ταλαιπωρίας των ζώων, η προστασία του περιβάλλοντος και τέτοια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη όταν εξετάζεται η κατοχήρωση ενός ζώου για δίπλωμα βιστεχνίας. Κύριε Ταραμπέλα, θα ήθελα να σας πω ότι πάνω από 20 χρόνια εργάζομαι στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και εξακολουθώ να ε, απολαμβάνω τη δουλειά μου και το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον και από κοινωνική και από δεοντολογική ηθική άποψη. Και πιστεύω ότι έχουμε εργαλεία για να δίνουμε σωστές λύσεις σε αυτά τα θέματα και εμείς στο γραφείο μας κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να ευθυγραμμιζόμαστε με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Μάλιστα. Τι να σας πω, μας αν θέλετε εσείς κόκκινα αγκούρια, τότε να κάνουμε τις ντομάτες πράσινες ή και μαύρες. Όλα είναι θέμα συνήθειας τελικά. Ο άνθρωπος συνηθίζει σε όλα. Σας ευχαριστούμε πάντως. Και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονες για την παρουσία σας. Γιατί καταφέρατε και κάνατε μία ανακεφαλαίωση και απαντήσατε συνοπτικά σε τόσο δύσκολες ερωτήσεις και μας δώσατε αρκετές εξηγήσει. Οι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, όπως του κυρίου Άγνιου και άλλων, ήταν τόσο ενδιαφέρουσες που μας έδωσαν τροφή για σκέψεις και όρεξη να επανέλθουμε στο θέμα αυτό σε άλλη ευκαιρία. Πάντως, πραγματικά καταφέρατε και μέσα σε λίγο χρόνο απαντήσατε σε πολλές ερωτήσεις. Θα προβλέψουμε και νέα δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων και μάλιστα σχετικά σύντομα. Οπότε η σημερινή μα συνάντηση σίγουρα δεν θα είναι τελευταία. Γιατί διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενημέρωσης για τα θέματα αυτά. Για να αντιληφθούμε καλύτερα τόσο περίπλοκες διαδικασίες. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις σχέση που έχετε με τις χώρες μέλη, αλλά τώρα δεν προλαβαίνω την επόμενη φορά. Σας ευχαριστούμε θερμά πάντως. Αλλά και μία ώρα να είχατε επιπλέον, πάλι δεν θα καταφέρατε να απαντήσετε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις και τις απορίες. Θα επανέλθουμε λοιπόν άλλη φορά. Ολοκληρώνουμε αυτό το θέμα. Έχουμε ένα τέταρτο για κάθε ένα από τα υπόλοιπα θέματα. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουμε με τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε το θέμα του γενικού προπολογισμού. Κύριε Σάνη, ένα τέταρτο μόνο μπορούμε να αφιερώσουμε στο θέμα σας. Το γενικό προπολογισμό δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018. Δεν θα σας ε, φάω χρόνο. Επί το έργο παρακαλώ, κύριε Σάνι, μόνο ένα τέταρτο έχουμε για τη συζήτηση αυτού του θέματος. Να τεθούν ερωτήσεις και να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Σάνη, παρακαλώ. Thank you uh, Ευχαριστώ, πολύ. Θα είμαι σύντομο. Μετά τον τριμερή διάλογο θα σα παρουσιάσω το σχέδιο νομοδότηση σε σχέση με τον ε, προπολογισμό. Όλοι συμφωνούμε για την σημασία τη γεωργία και τη ανάπτυξη ε, τη επέδοση των Υπάρχει λοιπόν και ενδιαφέρον από το γεωργικό τομέα για τον νέο προπολογισμό. Έχουμε νέα σημαντικά στοιχεία τα οποία βεβαίω θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να τονίσουμε μόνο κάποια συγκεκριμένα σημεία. Έχουμε ένα πολιετέ ε, πρόγραμμα και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στην επικεφαλίδα 2 ο προπολογισμό θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ή και ενδεχομένω θα αυξηθεί, συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών φακέλων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πέρα των επαναπληρωμών ε, λόγω παρατυπίων στη Γεωργία θα πρέπει να παραμείνει το θέμα αυτό στην επικεφαλίδα 2. Επίσης, οι δεσμεύσει για τις πληρωμές θα πρέπει να παραμείνουν στο πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ένα ιδιαίτερο σημείο αφορά το Brexit που θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Γεωργία μελλοντικά. Και καλούμε την Επιτροπή να λάβει υπόψη στον υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο. Επίση, θα πρέπει να σα αναφέρω ότι το 2018 θα έχουμε το τελευταίο έτσι, εύκολο δημοσιονομικό έτος, επειδή ακριβώς θα έχουμε τις νέες ε, τις νέες χρηματοοικονομικές, νέες δημοσιονομικές καταστάσεις μετά από αυτό το σενάριο. Θα πρέπει λοιπόν να επιδείξουμε ευθύνη σε σχέση με τον προπολογισμό τη ΚΑΠ τη στιγμή που υπάρχουν σοβαρέ απειλές όσον αφορά το ΠΔΠ. Θα πρέπει να είμαστε λογικοί και θα πρέπει να προσπιστούμε αυτό που έχουμε και θα πρέπει να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι συναδελφοί μας αναθέτοντά μου μάλιστα να ασχοληθούμε αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να, δι, ε, να διευκολύνουμε τη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τη ΚΑΠ. Θα πρέπει να δούμε ακριβώ τι θα γίνει και με το όμνιμπο στα πλαίσια του προπολισμού 18-19. Θα πρέπει να δούμε για τι που υποχρεώσεων τι γίνεται με την καταπολέμηση των ε, επιζωοτιών και τα 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πρέπει ενδεχομένως να αυξηθούν, επειδή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αύξηση αυτών των πιστοτήτων. Προπαρασκευαστικές δάσεις και επιπλέον προγράμματα θα πρέπει να αφορούν την αναπτύξη της υπέτρου. Προσβλέπω πάντως, ε, συνάδελφοι, στις τροπολογίες σας, στη συνεργασία με τους Κιώδης και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής και ήδη αυτό μου πήρε δύο λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μπράβο σα. Κυρία Μίλλερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την προκαταρκτική εργασία του εισηγητού, τον οποίο υποστηρίζουμε. Για μας είναι βέβαια επίκαιρο με το Brexit δεν πιέζει τόσο πολύ. Μας ενδιαφέρει περισσότερο το ρωσικό εμπάργκο Οι Βέλγοι συναδελφοί μου μου επισημαίνουν διαρκώς ότι δεν αντισταθμίζονται οι ζημίες τους, δεν ε, αποζημιώνονται. Στο, για το Omnibus έχουν ξεκινήσει τριμερείς διάλογοι, δεν ξέρω αν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον προπολογισμό του 2018, ούτε και το ρωσικό εμπάργκο άλλωστε. Γενικώ πάντω τασόμαστε υπέρ τη έρευνα, υπέρ τη αύξηση των κονδυλίων για την αντιμετώπιση των επιζώτιων. Εν τέλει είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εκθεσή σα και σα ευχαριστούμε για αυτήν. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο από την Ομίγυρη. Σα ευχαριστώ θερμότατα. Ο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ο κύριος Χόισλερ. Α, συγγνώμη, ξέχασα κάποιο συνάδελφο. Δεν βλέπω το όνομά σας από μακριά. Παρακαλώ. Έχω κάποια σχόλια για την έκθεση Σάνι. Ε, τα περισσότερα σχόλια είναι θετικά βέβαια, γιατί οι προ, προτάσεις ε, προ, προβλέπουν αντιστάθμιση του Brexit, ε, ε, χρηματοδότηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον επιστηστικό τομέα και επίσης εξασφάλιση χρηματοδότησης για τα πιλωτικά προγράμματα ώστε να αναχαιτιστεί η απερίμωση της υπαίθρου. Αυτά είναι τα θετικά. Το αρνητικό είναι ότι το βάρος του γεωργικού προϋπολογισμού ε, όλο και μειώνεται στο σύνολο του κοινοτικού προϋπολογισμού και είναι ακόμη το 38% του συνόλου του κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά φοβόμαστε περαιτέρω περικοπές. Και μάλιστα πολλοί συνάδελφοι θεωρούσαν ότι παρόλο που έχει μειωθεί ο γεωργικός προϋπολογισμός ε, εξακολουθεί να είναι υπέρογος. Η κοινή γεωρική πολιτική όμω είναι η μοναδική πανευρωπαϊκή πολιτική και η χρηματοδότησή τη αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό τη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να περικόψουμε περαιτέρω το προπολογισμό τη κοινή γεωρική πολιτική αν δεν προβλέψουμε ουσιαστικέ εναλλακτικέ λύσει που να ενισχύουν την επιστηστική κυριαρχία των λαών τη Ευρώπη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα προϊόντα μα αλλά και του παραγωγού μα, άνδρε και γυναίκε, απέναντι σε απειλέ που συνιστούν οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών, που θα αποδυναμώσουν ακόμη περισσότερο το ρόλο των απλών απέναντι στι πολυεθνικές και ο ρόλος ε, της ομάδας μας είναι πολύ σημαντικός και της Επιτροπής, γιατί βρισκόμαστε σε διαδικασία μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε άρδιν το γεωργικό και κτηνοτροφικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για να λάβει υπόψη την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία, αλλά για να περάσουμε από μια νοοτροπία της επιχορήγησης σε νοοτροπία προστασίας των δικαιωμάτων των χωρικών των αγροτών. Και ε, στη ε, μέση για τα προϊόντα που θα λαμβάνουν υπόψη και το περιβαλλοντικό κόστος και την ανθρώπινη υγεία. Γιατί για κάθε ευρώ που ξοδεύουμε σε προϊόντα της συμβατική γεωργίας και βιομηχανικής γεωργίας πληρώνουμε 2 ευρώ από την κοινωνία για τις ε, δαπάνες υγείας. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μαρτίνες και τώρα ο Διευθυντής, ο κύριος Χόισλερ. Παρακαλώ και εσείς ε, σύντομα. Thank Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Θα απαντήσω σε κάποια θέματα που τέθηκαν. Καταρχά, το Brexit. Ναι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν θα υπάρξει για το 2018 οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συνόμενο αντίκτυπο. Μετά θα αλλάξουν τα πράγματα. Να αφιστήσω την προσοχή σας επίσης την προσοχή στο θέμα των εισοδημάτων. Αναμένουμε την ομαλοποίηση των διαδικασιών, οπότε τα εισοδήματα από αυτή τη διαδικασία θα είναι πιο χαμηλά. Άμεσες πληρωμές. Νομίζω ότι τώρα είμαστε σε ταχύτητα πλεύσης, οπότε υπάρχει θετική εξέλιξη για αυτό το κομμάτι. Δύο λόγια και για τα μέτρα για τις αγορές. Είδατε ότι δεν προβλέπουμε πιστώσεις όσον αφορά τον τομέα της κτηνοτροφίας αυτή τη χρονική στιγμή. Υπάρχουν 71 εκατομμύρια για φρούτα και λαχανικά, αλλά βεβαίως η Κομισιόν θα συνεχίσει να επαγρύπνα αν χρειαστεί να παρενέβει στον τομέα της κτηνοτροφίας. το ΠΔΠ μας υποχρεώνει να παραμείνουμε στα κάτω από τα όρια. Καταρχάς έχουμε το απόθεμα για τις ε, κρίσεις, το οποίο θα ακολουθήσει στην συνδικασία όπως ξέρετε. Ανάπτυξη Πέθρου, εδώ έχουμε καλά νέα. Βρισκόμαστε σε πάλι ομαλή εξέλιξη όσον αφορά τις ε, προπληρωμές και νομίζω ότι εδώ τα πράγματα εξελίσσονται καλά. και να σας ευχαριστήσω επίσης και για τις προτάσεις για τα πιλωτικά προγράμματα. Νομίζω ότι η Κομισιόν έχει απαντήσει επισήμως και θα περάσουμε τώρα στις ε, διαπραγματεύσεις με εσάς. Πάντως, να σας πω διαδικαστικά ότι θα λάβετε μια τροποποιητική επιστολή το φθινόπωρο που θα λαμβάνει υπόψη της τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την εκτέλεση των άμεσων πληρωμών. Όπως ξέρετε, τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα τα τέλη του Οκτώβρη και θα είναι τμήμα της συνδιαλλαγής. Και καταλήγοντας, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επαναφορά των κονδυλίων που προτείνει η Κομισιόν. Επειδή ξέρετε ότι το Συμβούλιο θα έχει αντίστοιχη θέση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ο κύριος Αντριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιγραμματικά θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα των πιλωτικών προγραμμάτων. Είναι σημαντικά. Θα πρέπει πρώτα να αποφύγουμε την, ε, την υποβάθμιση των ε, αμπελιών γιατί η αμπελουργία έχει μεγάλη σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έρευνες, ε, ειδικέ έρευνες στον αμπελουργικό τομέα. Το θέμα αφορά όλα τα αμπέλια, γιατί είχαμε ε, φιλοξήρα στην αρχή του αιώνα, αλλά έχουμε εξίσου δραματική περίπτωση και τώρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αμπέλια μας ε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το λόγο έχει και πάλι ο εισηγητής ο κύριος Σάνη. Ευχαριστώ. Αυτά. Μάλιστα, 14 Ιουλίου λίγη διορία για την υποβολή τροπολογιών στη μία το μεσημέρι. και έχουμε τη σχετική έγκριση των συντονιστών. Περνάμε στο επόμενο θέμα, την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της, του κατεξοδότηση κανονισμού που τροποποιεί το κανονισμό 697 του 2009 για τις αμπελονικές ποικιλίε στα συνώνυμά τους που εμφανίζονται σε ετικέτες κρασιού. Έχουμε τον κύριο Ζωάνο Νοφρέ από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη που ασχολείται με το τμήμα κρασιών αλκοολοχών ποτών και ειδικών καλλιεργιών και προϊόντων. Στις 19 Μαΐου ε, είχαμε τον κανονισμό που τροποποιούσε το κανονισμό 607-219 για τις αμπελονικές ποικιλίε και τα συνώνυμά τους που μπορούν να εμφανίζονται σε τικέτες ίνου. Ε, μάλιστα με προθεσμία για υποβολή αντιρρήσεων την 19η Ιουλίου του 2017 υπευλήθη από τον κύριο Φρανκ Μπόκοβιτς ε, Σλοβαίνο του ΕΛΚ έτοιμα για παράταση της ε, προθεσμίας αυτής κατά δύο μήνες. Στην κατεξοδότηση πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τροποποιήσει τον κανονισμό ώστε να επιτρέψει και στους ε, Κροάτες Ινοπαραγωγούς να περιλαμβάνουν στην προστατευόμενη ονομασία προέλευση, προέλευσης Κροατική Ίστρια και τον όρο Τεράν για την ε, ποικιλία κρασιού. Τέτοια ποικιλία με το ίδιο όνομα ήδη καλύπτεται από τη σλοβενική προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Θα μας ε, διευκρινίσει καλύτερα την κατάσταση βέβαια ο αρμόδιος ε, διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη, ο κύριος Ονοφρέ. Ξέρω ότι το σύστημα είναι περίπλοκο και μακάρι να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο. Και νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν είχαμε μια γευσηγνωσία, έτσι θα καταλαβαίναμε καλύτερα τις διαφορές. Εν πάση περιπτώσει έχετε μόνο λίγο χρόνο, 10 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να καταφέρω να διασκεδάσω τις ανησυχίες σας και να διευκρινίσω ε, τις αφιβολίες που έχετε. Χαίρομαι για την ευκαιρία που μας ε, δίνετε να σας παρουσιάσουμε για πρώτη φορά τις απόψεις μας για την κατεξοδότηση πράξη. Το θέμα αυτό συζητήθηκε επανειλημμένως στην Μόνιμη Επιτροπή Γεωργίας και στο Συμβούλιο, αλλά για πρώτη φορά εγκύπτει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν, αντίθετα με ό,τι εσφαλμένως ισχυρίστηκαν πολύ ενδιαφερόμενοι, δεν αφορά αυτή η κατεξοδότηση πράξη μόνο δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατεξοδότηση πράξη αφορά μία εξαίρεση από το, τους γενικούς κανόνες ετικετοθεσίας του ίνου και την υιοθέτηση μιας εξαίρεσης για τους κανόνες αυτού. Οι γενικοί κανόνες για τη σήμανση του ίνου δεν επιτρέπουν τη χρήση ονόματος μιας εμπελονικής ποικιλία όταν ε, περιέχει η, αποτελεί την, μια προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Με την εξαίρεση αυτή όμως, ε, μάλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαιούται αν πληρούνται δύο προϋποθέσεις, να προβλέψει εξαίρεση με καταξιοδότηση πράξη. Ποιε είναι οι δύο προϋποθέσεις. Καταρχήν, το όνομα αυτό, απόδειξη τέτοιου ονόματος για την προστατευόμενη νομασία προέλευση και προϋπάρχουσες πρακτικές σε σχέση με αυτή την αμπελονική ε, ποικιλία. Οι δύο αυτές προϋποθέσεις συντρέχουν πλήρω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 53 ε, παρόμοιες εξαιρέσεις ε, από την αμπελοϊνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ωφελούν όλα τα αμπελοϊνικά κράτη-μέλη, κυρίως τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, ακόμη και τις κάτω χώρες. Όλες, όλες οι χώρες που παράγουν ίνο εποφελούνται από τέτοιες εξαιρέσεις. Γιατί λοιπόν να έχουμε διαφορετική μεταχείριση στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν μια ε, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης προστατεύεται και μία ανώνυμη, ανώνυμη ποικιλία χρησιμοποιείται για αντίστοιχη προστατευμένη ε, ονομασία σε άλλη χώρα. Άλλωστε δεν γίνεται καμία παραπλάνηση του καταναλωτή. Ισχύει ότι και στις προηγούμενες εξαιρέσεις. Και για λόγους ίση μεταχείριση των κρατών μελών και οι Κροάτες παραγωγή θα πρέπει να υποφεληθούν αυτής της εξαίρεσης και να γίνει ε, να διεκπαιρεωθεί αυτή η κατεξιοδότηση. Επίσης δεν επηρεάζονται οι Σλοβαίνοι παραγωγή του ίνου Τεράν, γιατί ε, κρατούν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και το Τεράν είναι μια αποκλειστικώς σλοβενική προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Αλλά με τη συγκεκριμένη κατεξοδότηση πράξη προβλέπουμε καλύτερη προστασία της ΠΟΠ Τεράν, γιατί περιλαμβάνει μία μοναδική προστασία με το μέγεθος των χαρακτήρων, ώστε να αποφευθεί παραπλάνηση του καταναλωτή. Έτσι, οι σλοβενικές και Κορατικές αρχές ε, είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν ώστε να αποτρέψουν πιθανές καταχρήσεις ε, στην επισήμανση αυτού του ίνου. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ένα κατάλογο μιλητών που δήλωσαν επιθυμία να λάβουν το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ενάμιση το πολύ. Η κυρία Πετήρ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την εισαγωγή. Θα ήθελα να πω ότι είμαι κατά οποιασδήποτε παράταση της προθεσμίας για να ε, καθυστερήσει η εφαρμογή αυτής της κατεξοδότησης πράξης. Νομίζω ότι ήταν ε, το μόνο που μπορούσε να κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υιοθετήσει κατεξοδότηση πράξη, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις. Και μάλιστα έχουμε μια σειρά εξαιρέσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επιτρέπεται η δυνατότητα ε, τίτλου ε, ονομασίας ομπελονικής ποικιλία και σε περίπτωση ε, προστασίας ε, ονομασίας προέλευσης. Έχουμε μία ακόμη προστασία για το τεράν που προστίθεται στις 53 εξαιρέσεις που ήδη ισχύουν. Έχουμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία αντίστοιχες περιπτώσεις. Είναι απαράδεκτη η στάση της Σλοβενίας που δεν θέλει να επιτρέψει για την Κροατία κάτι που ε, ίσχυσε για την ίδια και από το οποίο υποφελείται η ίδια. Ήδη έχουμε μία τριετία που περιμένουν ε, οι Κροάτες παραγωγοί σε δυσμενή θέση να υιοθετηθεί αυτή η κατεξοδότηση πράξη και έχουν υποστεί πολλές οικονομικές ζημιές. Είναι ανεδαφικά τα επιχειρήματα της Σλοβενίας για την παράταση της προθεσμίας. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις, πληρούνται οι... τα σχετικά άρθρα. Ζητήσαμε εξαίρεση για να περιληφθούν ε, στον τίτλο και ε, όρος τεράν ε, αμπελονική ποικιλία με, στα κρασιά που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης Κροατική Ίστρια. Νομίζω ότι συντρέχουν όλε οι προποθέσει και δεν έχει νόημα το αίτημα τη Σλοβενίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόγκοβιτ. First of all, I protest because I cannot... Διαμαρτύρομαι πρώτα διότι δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα την ζήτησα αλλά δεν μου επέτραπη. Ε, ύστερα θέλω περισσότερο από ένα λεπτό για να, για να εξηγήσω. Πρώτα, Τεράν είναι προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ενός κρασιού που προέρχεται από ποικιλία κρασιών που καλλιεργείται στην περιοχή κράση. Η ειδική περιοχή για πρώτη φορά προστατεύθηκε από το από τα 1917 στην ε, πρώην Ιουγκοσλαβία. Και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προστατεύεται και έχει καταχωριστεί ως προστατευόμενη ονομασία από τις 17 Φεβρουαρίου 2006. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κάθε χώρα μέλος ή τρίτη χώρα η τρίτη χώρα ξαναλέγω που επιθυμεί να παράγει κρασί με την ίδια ονομασία που περιλαμβάνει ωστόσο ποικιλία με προστατευόμενη ονομασία, οφείλει να ζητήσει εξαίρεση όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τέτοια αίτηση μπορεί να γίνει. Ενδεχομένω σε ενταξιακέ διαπραγματεύσει για να υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα σε περίπτωση ήδη προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Κροατία δεν ζήτησε η ποικιλία κρασιού που ονομάζεται Τεράν να περιληφθεί στην λίστα των εξαιρέσεων όπως είχε κάνει για ορισμένε άλλες ποικιλίε κρασιών. Κάτι έγινε μετά όμως πραγματικά ασυνήθιστο όπως διαβάζουμε στην ε, στην πράξη υποσχέθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά μετά από την ένταξη της χώρας αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εφόσον η Σλοβενία θα παρατείται από την προστασία του δικού της ε, κρασιού. Με αυτή την πράξη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη στην προστασία της γραφικής ένδειξης του κρασιού αυτού και μάλιστα νομιμοποίησε την υφιστάμενη παράνομη πρακτική επισήμανσης ε, προϊόντων και επομένως παραβίασε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, ανοίγουμε εδώ την πηξίδα της Πανδώρας σε ό,τι αφορά την καταχώρηση προστατευόμενων ε, ενδείξεων προέλευσης αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αύριο, αγαπητοί μου Ούγγροι συνάδελφοι, μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια στην πράξη με εξαίρεση για την ε, κατάρχηση προστασία του Τοκάι. Κάποιο μπορεί να εμφανιστεί με την ιδέα ότι το ιταλικό κρασί Μπαρόλο, προστατευόμενη ονομασία στην Ιταλία, ιδίω στην περιοχή Πιεμόντε, ε, δεν θα προστατεύεται επαρκώς. Θέλουν να χρησιμοποιήσουν άλλη την ονομασία αυτή, να την βάλουν πάνω στα μπουκάλια του κρασιού που παράγουν. Αυτά είναι αναπαράδεκτα πράγματα. Είμαι πεισμένο ότι η στην πράξη θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν για την εξαίρεση για την επισήμανση κρασιών. Για αυτό το λόγο σας ζητώ εξ ονόματος των Σλοβαίνων παραγωγών κρασιού Τεράν να εγκρίνετε δίμηνη παράταση στην προστασία. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές, θα ήθελα να πω στην κυρία Πέτυρ ότι έχει δυνατότητα και συμπληρωματικού χρόνου γιατί ο κύριος Μπόκοβιτς μακρηγόρησε, οπότε και εσείς δικαιούστε να μιλήσετε και λίγο παραπάνω, αν επιθυμείτε να επανέλθετε. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, και μετά την παρουσίαση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η κατεξοδότηση πράξη επιτρέπει στην Κροατία να εμπορευτεί ε, κρασιά με το όνομα Τεράν ε, κρασιά που έχουν προστατευόμενη ονομασία προέλευση στην κροατική ύστρα. Και μάλιστα χρησιμοποιεί τον όρο ταράνι και που χρειάζεται. Μάλιστα ήδη τέσσερα χρόνια καθυστερεί η εφαρμογή αυτή τη απόφαση. Στο μεταξύ, οι Κροάτε παραγωγοί είναι σε δυσμενή θέση σε σχέση με του υπόλοιπου και έχουν υποστεί ανεπανόρθωτε και αδικαιολόγητε οικονομικέ ζημιέ. Η Κροατία έχει εκπληρώσει τι προποθέσει ε, για την ισχύ τη εξαίρεση με βάση την κοινωτική νομοθεσία. Ε, κάτι που συνδέεται άμεσα με την ε, υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει προστατευόμενη νομασία προέλευση με την ένταξη τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει λόγο για να καθυστερήσει περαιτέρω η θέση σε εφαρμογή τη κατεξόδηση πράξη, προκειμένου ε, τα κρασιά της ε, POP ΠΟΠ Κροατική Ίστρα να περιλαμβάνουν ως τίτλο το «Την ποικιλία Τεράν» η παράταση μόνο στρέβλωση ανταγωνισμού συνιστά. Γι' αυτό σας ζητώ θερμά να καταψηφίσετε το αίτημα για αναβολή της α, θέσης ισχύ της α, πράξης για ένα δίμηνο ακόμη. Ευχαριστώ κύριος Γιακόφτσης. Είναι αλήθεια ότι εδώ και 800 χρόνια παράγεται στην Ίστρια το κρασί τεράν. Είναι αλήθεια ότι για το κόκκινο κρασί και για τους ε, κατοίκους της Ίστρια το τεράν είναι συνώνυμο του κόκκινου κρασιού. 800 χρόνια παράγουμε ένα κρασί που ε, εξυπηρέτησε και την ε, Αυστρογγρική αυλή ένα διάστημα. Είναι απόδειξη ότι έχουμε μακραίωνη παράδοση παραγωγής του Ίνου Τεράν. Εμεί δεν θέλουμε να σφετεριστούμε το δικαίωμα κανενό. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικά μα δικαιώματα. Και είμαστε αν, αν, είστε λοιπόν υπέρ τη βιοπικιλότητας, υπέρ τη προάσπιση τη πολιτιστική και τη περιφερειακή ταυτότητας, υπέρ των ντόπιων προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωση. και αν είστε υπέρ του σεβασμού των ε, αρχών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσετε κατά ε, κατά της παράτασης της προθεσμίας, γιατί αυτή η δίμηνη παράταση της ε, θέση ισχύ της κατεξόδησης πράξης δεν πρόκειται να λύσει τίποτα. Εδώ και 5-6 χρόνια προσπαθούμε με τους Σλοβαίνους να βρούμε κοινή λύση. Εγώ πρότεινα λύση για διασυνοριακή και να χρησιμοποιηθεί όρος Τεράν, γιατί Τεράν, κρασί, δεν παράγεται μόνο στη Σλοβενία και στην Κρόατια, αλλά και στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά δεν έγινε δεκτή ούτε μία πρόταση από τους Σλοβαίνους συναδέλφους. Είναι λοιπόν καιρός ε, να λάβουμε μία απόφαση. Ο χρόνος έχει περάσει, τέλειωσε η προθεσμία, είμαστε κατά της παράτασης προθεσμίας, θα πρέπει να δεθεί το συντομότερο δυνατό σε εφαρμογή η κατεξοδότηση πράξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία παράταση δεν πρόκειται να δώσει λύση, απλώς θα επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Ευχαριστώ. Ψηφίστε κατά. Σας ευχαριστώ κύριο Δες. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Ως συντονιστής της πολιτικής μου ομάδας θέλω να πω ότι εμείς έχουμε εγκρίνει την ε, λεγόμενη free vote, δηλαδή ψήφο κατά συνείδηση. Ο καθένας θα ε, αποφασίσει, θα ψηφίσει όπως επιθυμεί, δεν θα δώσω γραμμή. Ωστόσο, όσο καιρό είμαι συντονιστής Πρώτη φορά επιτρέπω τόσο μεγάλη ελευθερία ψήφου. Ορισμένοι εινοπαραγωγοί, πάντως ε, Γερμανοί εινοπαραγωγοί, με παρακάλεσαν να μην υπερψηφίσουμε την ε, παράταση, διότι και αυτοί αναμένουν να υποφεληθούν. Υπάρχει πλήθος ε, ρυθμίσεων, δεν θέλουμε αυτές οι εξαιρέσεις ε, των ρυθμίσεων να αμφισβητηθούν. Αυτό είναι, αυτό το νόημα της ε, ε, παράκλησής τους. Μάλιστα, δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Εκτός και κάποιος ξέχασε να ζητήσει το λόγο. Η κυρία Μαγκίνες, παρακαλώ. Πρόεδρε, να πω μόνο ότι είναι αδύνατο να κάνουμε απόφαση, εκτός και αν έχουμε δείγματα του κρασιού για να δοκιμάσουν συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, τώρα κατάλαβα γιατί συγκεντρώσατε τόσες ψήφους στην εκλογή σας στη θέση του Αντιπροέδρου. Πάντως η ιδέα σας πραγματικά ήταν φαϊνή. Εγώ το είπα με πιο διακριτικό τρόπο, δεν τόλμησα να το πω τόσο ξεκάθαρο όπως εσείς, τόσο σταράτα. Εν πάση περιπτώσει, ας περάσουμε στην ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε επί του αιτήματο παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της αντίρρησης. Αν εγκριθεί το αίτημα, τότε θα παραταθεί μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνω. Ε, παρατείνεται, αν εγκρίνουμε το αίτημα, για ένα δίμηνο την προθεσμία για την υποβολή έστασης. Μέχρι τις 19 ε, Σεπτεμβρίου θα παραταθεί η προθεσμία για την υποβολή έσταση σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για παράταση. Έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες, παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Α, κατέφτασε η κυρία Σένερα. Proszę mi wybaczyć. να με συμπαθάτε. Τέλος ψηφοφορίας. 5 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται το αίτημα παράταση προθεσμίας. Δεν πρόκειται λοιπόν να παραταθεί μέχρι το Σεπτέμβριο η σχετική προθεσμία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Έχουμε ακόμη ένα σημείο, το τελευταίο, έγκριση των συστάσεων των συντονιστών τη Επιτροπή Γεωργία. Σας έχουμε στείλει ηλεκτρονικά τις αποφάσεις των συντονιστών, αλλά και γραπτός. Αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις ή αντιρρήσει, επιβεβαιώνονται οι συστάσει των συντονιστών. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι την τελευταία μας συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές. Σας εύχομαι θερμότατα καλές διακοπές. Μας περιμένει πολύ έντονο φθινόπορο. Γι' αυτό ξεκουραστείτε για να μου έρθετε ακμαίοι το φθινόπορο. Ευχαριστώ θερμά και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους και στους διερμηνείς. Λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε και νωρίτερα μάλιστα λίγο. Ευχαριστώ και πάλι σας ευχαριστώ όλους θερμά. Λύεται η συνεδρία της Επιτροπής Γεωργίας.